Ladies and gentlemen, shall we Μπορούμε να ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε... Έχουμε ήδη, έχει ήδη περάσει ένα τέταρτο και έχουμε 32 σημεία στην ημερήσια διάταξη. 32. Ας περάσουμε λοιπόν στην έγκριση του σχέδιου ημερήσιας διάταξης. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν αντιρρήσεις. Ναι, κύριε Πρόεδρε, εάν στην συνεδρίαση των συντονιστών ληφθεί απόφαση επί της διαδικασίας, ιδίως για το Πακιστάν, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε νωρίς το μεσημέρι. Να δούμε πώς μπορούμε να το βάλουμε στη διάταξη. Ναι. Καθίστε πρώτα να δούμε αν θα υπάρξει απόφαση. Μπεν Λάγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σε σχέση με, μια, σε σχέση με την απόφαση των συντονιστών βεβαίως, αλλά θεωρώ ότι θα είναι θετική έκβαση. Θα παρακαλούσα στο σημείο ψηφοφορία να συμπεριληφθεί και η ψηφοφορία για ένα προφορικό ερώτημα σε σχέση με την Κολομβία. Γιατί συζητήσαμε και συμφωνήσαμε με τις πολιτικές ομάδες, ούτως ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί συνοδευτικά ε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Περού και την Κολομβία. Να υποβληθεί δηλαδή αυτή η προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν. Ε, Περνάμε στο σημείο 2, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας του Μαρτίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις πριν το τέλος της συνεδρίασης, όσοι ήθιστε θα θεωρηθούν ότι εγκρίνονται όπως ε, ήθιστε επίσης ε, μεταδίδεται στο δίκτυο, στο διαδίκτυο η συνεδρίαση μας πλην βέβαια τη συνεδρίαση κυκλισμένων των θύρων. Η λίστα του βιβλιογραφίας έχει διανεμηθεί. Αν σας ενδιαφέρει κάτι ζητήστε το παρακαλώ. Σημείο 4. Πρόοδος των τριμερών διαπραγματεύσεων. Έχουμε δύο ε, φακέλους που διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο Διμερείς Επενδύσεις, Συμφωνίες, Συνθήκες. Και θα σας πω πώς έχει κατάσταση. Έχουμε συμφωνήσει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να διαμεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας. Η Κομισιόν Έχει λοιπόν παρουσιάσει ένα ανεπίσημο έγγραφο non-paper και πλέον το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει αν συμφωνεί με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και από πλευράς μας θα πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς εάν δεχόμαστε αυτό το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακόμη πετύχει τη συμφωνία. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο θέματα, τα οποία πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Την επόμενη όμως εβδομάδα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα γνωρίζουμε κατά πόσον θα έχουμε συμφωνία ή όχι τελικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον οργανισμό GSP, έχει ξεκινήσει ο τρομερής διάλογος. Όπως ξέρετε, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια, αλλά να ξεκινήσουμε άμεσα και τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ο συγητής μας, κύριος Φιέλνερ, θα μας ενημερώσει σχετικά. I think we've made a lot of way actually uh, in this file and uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε κάνει πρόοδο. Και αυτό γιατί ακόμη και πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ήταν σαφές ότι το Συμβούλιο δεχόταν σε μεγάλο βαθμό το συμβιβασμό που είχαμε εμεί εδώ στο Κοινοβούλιο εγκρίνει. Αυτό ήταν λοιπόν ένα θετικό σημείο εκκίνηση. Στο χθεσινό τριμερή διάλογο ουσιαστικά διευθετήσαμε όλα τα τεχνικά ζητήματα και τα λιγότερο λεπτά από πολιτικής πλευράς ζητήματα. Και τώρα αυτό που μένει ουσιαστικά είναι αν θέλετε η ουσία τα πραγματικά ευαίσθητα λεπτά ζητήματα έχουν μείνει. Τέσσερις τομείς κυρίως, ασφαλιστικές δικλίδες, διάρκεια, προϊόντα και κάποιες ε, αρχές σχετικά με τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Εμείς ως Κοινοβούλιο κάναμε την προσφορά μας προς το Συμβούλιο και περιμένουμε την απάντησή τους για ένα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο φάκελο. Αλλά το κλίμα είναι πολύ καλό και επειδή και τα δύο θεσμικά όργανα πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά δεν έχουμε κάνει ακόμη τα βήματά μας δεν έχουν ακόμη ας πούμε ευθυγραμμιστεί, αλλά πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και νομίζω ότι πριν τη δεύτερη ολομέλεια του Μαΐου θα έχουμε καταλήξει έτσι θα σφραγίσουμε επί της Δανικής Προεδρίας μάλλον ε, την συμφωνία. Ευχαριστώ. Επιτρέψατε μου να αναφερθώ σε εξή θέματα. Καταρχήν την ομάδα διαπραγμάτευσης στο Κοινοβούλιο έδειξε πραγματικά αξιοσημείωτη ενότητα στη Σπήρωση και αυτό είναι πολύ καλό όσον αφορά τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να μοχλεύσει τη διαπραγματευτική του ικανότητα με το Συμβούλιο. Τώρα θα περάσουμε στο σημείο 4 τη πρόοδο των τριμερών διαπραγματεύσεων και θα κάνω κάποιες σύντομες αναγγελίες ως προς την κατάσταση εκτός βεβαίω από εκείνα τα θέματα που δεν έχουν σημειωθεί εξελίξεις. Ξεκινώντας με την ε, Ρωσία, ε, Κύριε Πρόεδρε, ε, προσπαθήσαμε να έχουμε μια συνάντηση με τον Ρώσο πρέσβη και δυστυχώς είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε μια ημερομηνία που να μπορεί να συναντηθεί μαζί μας. Περιμένουμε την πρώτη συνάντηση, μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Επιπρόσθετα προς τις ε, πληροφορίες που δώσαμε στην τελευταία συνάντηση, θα ήθελα να πω ότι προετοιμάζουμε μια βραχία συνάντηση με την Επιτροπή όσον αφορά την ε, κατάσταση των επενδύσεων, της συνθήκης για τις επενδύσεις. Μετά από τις δύο πρώτες ανταλλαγές, μία με την Επιτροπή και τη Γενική Κατάσταση των Εμπερικών Σχέσεων και κατά δεύτερο λόγο με τον Πρέσβη, θα εστιάσουμε στην Συμφωνία Συνθήκη για τις Επενδύσεις. Τώρα Λοιπόν, θα ακολουθήσει ε, μια σημαντική συνάντηση με την κυρία Σπύρο, που είναι η εκπρόσωπος ε, της ε, Ευρώπης και ένα από τα βασικά θέματα θα είναι οι εξελίξεις για την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ευρω... Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Για τώρα για την Ιαπωνία. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την ομάδα παρακολούθησης για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας έγιναν τρεις συναντήσεις. Η ομάδα παρακολούθησης συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, το Συμβούλιο Επιχειρής της Ευρώπης στην Ιαπωνία και είχαμε και μία σύντομη συνάντηση με τον ε, Δανό πρέσβη υπό την της Ανικής ε, Προεδρίας και λίγο πολύ το επίπεδο των συζητήσεων σε σχέση με τα scoping exercises ε, συνεχίζονται. Δηλαδή, στις αρχές Μαΐου θα υπάρξει η τρίτη συνάντηση αυτής της ομάδας που θα προσπαθήσει να άρει τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμα σε σχέση με τον ορισμό αυτού του scoping exercise. Euh, και ελπίζουμε ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου θα καταλήξουμε σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό, ούτω ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε εκ μέρου τη Επιτροπή στο Συμβούλιο να οριστεί ένα πλαίσιο έναρξη των διαπραγματεύσεων, μια σχετική εντολή. Ακολουθούμε λοιπόν τι εξελίξει εκ του σύνεγγε και, εν πάση περιπτώσει, αύριο θα έχουμε τη συζήτηση με τον πρέσβη τη Ιαπωνία και πιστεύω ότι θα έχουμε επίσης τη δυνατότητα να του περάσουμε ξεκάθαρα το μήνυμά μας, δηλαδή τις προσδοκίε μας, να κάνει ό,τι μπορεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω να ακούσουμε τον πρέσβη της Ιαπωνίας και την, την Επιτροπή. Ζητήσατε το λόγο. Ε, ναι, Πρόεδρε. Εγώ για τη Μερκοσούρο. Γίνανε δύο συναντήσεις. Η μία ήταν ε, ε, χτες. πρόκειται για διαπραγματεύσεις εξαιρετικά δύσκολες και ευαίσθητες που συνεχίζονται. Γίνανε κάποια βήματα μπροστά, όχι πάντοτε γραμμικά, αλλά μπας περιπτώσει υπάρχει το θέμα της γεωργίας, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν ε, την εσωτερική αγορά του Μερκοσούρ, τις σχέσεις ανάμεσα στα διαφορά κράτη, ε, τις ε, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τη γραφειοκρατία, τη την βιομηχανία. Ακόμα δεν έχουμε περάσει σε ανταλλαγή προσφορών, γιατί η αντιπροσωπεία Μερκοσούρ δεν, δεν μας είπε ότι δεν μπορεί ακόμα να μας παρουσιάσει κάποια προσφορά. Γίναν κάποια βήματα μπροστά τόσο στην ομάδα για τους ε, κανόνες προέλευσης όσο και για την ειρηνική επίλυση διαφορών και για τη γεωργία. Εξετάστηκαν τα θέματα που σχετίζονται με τα φυτοϊγειονομικά ε, θέματα με τη λογική να φτάσουμε σε ομοιογενείς κανόνες σε ολόκληρη την Μερκοσούρ. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό ζήτημα το οποίο βαραίνει το Μερκοσούρ, για το οποίο, το, το οποίο μας ε, επηρέασε και την προηγούμενη εβδομάδα όταν συζητήσαμε το θέμα του Ρέψολ, το θέμα της σχέσης της Αργεντινής με τον υπόλοιπο κόσμο και πιο συγκεκριμένα με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για υποθέσεις όπως η Ρέψολ που είναι ο τελευταίος κρίκος μιας μακράς αλυσίδας. Ελπίζουμε ότι με την Βραζιλιάνικη Προεδρία που είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις ακόμα και με τη στήριξη της Ουρουγουάης και της Παραγουάης θα μπορέσουν να βελτιωθούν αυτά τα συστήματα σχέσεων με την Αργεντινή. Είναι ένα πρόβλημα που μας αφορά, αλλά αφορά κυρίως τον δικό τους τρόπο συμβίωσης μέσα στο πλαίσιο της ε, διάστασης της Μερκοσούρ. Ρωτήσαμε χθε αν ήταν δυνατόν να έχουμε μια επαφή με τον ε, πρέσβη της Αργεντινής. Ο πρέσβης μας απάντησε ότι δεν θα μπορέσει να μας ευχαριστήσει. Βάση περιπτώσει είναι μια από τις πιο σημαντικές ε, συμφωνίες που θα ήθελε να μπορέσει να ολοκληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά περισσότερο είναι πολιτική φύση η δυσκολία και όχι τεχνική, αν και στο θέμα τη Γεωργία εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τεχνική φύση και αντίθετα συμφέροντα. Έχουμε λοιπόν μεγάλε δυσκολίε, ωστόσο οι διαπραγματεύσει συνεχίζονται. Ο επόμενο διαπραγματευτικό γύρο θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Ήλιου και αμοιβαία μα ελπίδα είναι ότι η Βραζιλιάνικη Προεδρία θα μπορέσει να δώσει μια μεγαλύτερη όθεση προς μια... ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πίτερ είναι πολύ σύντομα για τον Καναδά. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I apologize, I just arrived, but I, I know it's, it's on the schedule. I was a little late. Uh. Ζητώ συγγνώμη που άργησα λιγάκι. Ε, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι Μόλις πριν ε, το Πασχαλινές Διακοπές είχαμε μια ομάδα παρακολούθησης εξαιρετική Εκτός από τη συμμετοχή του συναδέλφου είχαμε τους επικεφαλείς διαπραγματευτές, τον κύριο Πετροτσιάνα και τον κύριο Φερέλ. Ε, δίρκησε 45 λεπτά, το πίεσα όσο μπορούσα γιατί ήμουν μόνος που έθετε ερωτήσεις. Αλλά νομίζω πως μια από τις παρατηρήσεις μου συνεψίζει το τι συνέβαινε με κυρίως ο κύριος Βουέρχολ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής ε, του Καναδά, έκανε αυτή την εισαγωγική παρουσίαση για περίπου 10 λεπτά και μετά από λίγες ερωτήσεις και μετά μάλλον υποβλήθηκαν κάποιες ερωτήσεις. Ε, και μετά δεν ε, θεώρησα ότι έγινα πιο έξυπνος από ό,τι πριν, ότι κατάλαβα περισσότερα πράγματα από ό,τι πριν. Πάντως το θέμα είναι ότι τώρα η ομάδα σημείωσε πρόοδο Υπάρχει διαρκής πρόοδος. Τώρα ελπίζουν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το καλοκαίρι, ε, πριν το καλοκαίρι. Ναι, σε λίγες μέρες θα μεταβώ στον Καναδά. Σωθήκαμε. Φαίνεται να υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες, αλλά εν γέννη η επαρχία του Κουεμπέκ είναι υπέρ της συμφωνίας ΣΕΤΑ. Όπως, όπως και εγώ, όλοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τη μυστικότητα. Γι' αυτό όμως ονομάζεται C, comprehensive, ολοκληρωτική, δηλαδή όλα ή τίποτα είναι ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισαν να διαπραγματευτούν εμείς. Θα παρακολουθούμε, θα ακούμε ό,τι συμβαίνει. Τώρα μπορώ μόνο να εκφράσω την προσωπική μου ικανοποίηση, την δική μου αίσθηση, το τι αποκόμισα από τις ε, διαπραγματεύσεις με τους ε, επικεφαλείς ότι τα πράγματα δηλαδή προχωρούν σωστά και ότι θα ε, ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις εγκαίρω. Μάλιστα, ευχαριστώ. Εκουαδόρ, Βολιβία. Charles Σόλτς. Σόλτς. Thank you, Chair. I would ask, first of all, if we could agree that we are joining Bolivia and Ecuador in one monitoring group. Συμφωνήσαμε να τα βάλουμε την Βολιβία και το Εκουαδόρ. Να τους βάλουμε σε μία ομάδα παρακολούθησης. για το Εκουαντόρ, μετά από την εναρκτήρια σύσκεψη στη μέσα Μαΐου στην επόμενη συνεδρίαση θα ακούσουμε την Κομισιόν για το πεδίο τη προσπάθεια που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα για την πιθανότητα ε, ε, επανέναρξης διαπραγματεύσεων, ουσιαστικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ένωση και το Εκουαντόρ και έτσι να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιες είναι οι θέσεις των δύο πλευρών. Θα ακούσουμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση την επόμενη εβδομάδα και τότε θα σας ενημερώσω για αυτή την προσπάθεια στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ομάδες παρακολούθησης, για τους μόνιμους εξηγητέ που δεν είναι εδώ. Έχω κάποιες σημειώσεις για την Ινδία. Είχαμε μια επαφή με τον επικεφαλής διαπραγματευτή για τα εμπορικά θέματα μετά από τη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδία, για την Κεντρική Αμερική υπήρξε μια σύσκεψη με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και με τις ΣΜΚΟ και μου είπαν, αλλά δεν μπόρεσα να το επιβεβαιώσω, ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να χωρίσει το εμπορικό τμήμα αυτής της συμφωνίας, να το υπογράψει και να το θέσει σε προσωρινή εφαρμογή. Υπάρχει δηλαδή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μέσα στη συμφωνία σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική. Ουκρανία έγινε μια συνεδρίαση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελικά Σιγκαπούρη ε, συνεδρίαση με τους επικεφαλείς ε, διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε στη κοινή συζήτηση και, σημεία 6 και 7. Κοινή συζήτηση για την Κεντρική Αμερική. Πρώτα, Εμπορικός πυλώνας της συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών από τη μια πλευρά και Κεντρικής Αμερικής από την άλλη. Ο η συγκητής μα είναι ο Παύλο Φάλτα, αλλά θα αντικατασταθεί από την Μαρία Κορέια και Πρόκειται για τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Όπω γνωρίζετε, υπεύθυνο για την συγκατάθεση είναι η ΑΦΕΤ. Έτσι αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων ενάντια στη δική μας βούληση και στο δικαίωμά μας. Και Και μετά έχουμε τη διμερή ρήτρα για αυτή την εμπορική συμφωνία. Εμείς είμαστε λοιπόν εδώ υπεύθυνοι, αρμόδιοι και ήδη εξετάζουμε τις τροπολογίες στην έκθεση του. Δίνω το λόγο στους εισηγητές. Λοιπόν, πρώτα η Μαρία Κορέα. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας πω εξ ονόματος του συναδέλφου Παδός ε, Αλβάρο, ο οποίο ότι δεν μπόρεσε να έρθει εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου για να ασχοληθεί με τα εξή θέματα. Καταρχήν με τη Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ Κεντρική Αμερική και Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ρήτρα ε, διαφύλαξη ε, για να... της ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης. Καταρχήν θα ήθελα να εξάρω το πνεύμα αυτής της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου να παραμείνει ενεργή στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, σχετίζοντας αυτή τη Συμφωνία Σύνδεση με την Κεντρική Αμερική. Πρόκειται για μια συμφωνία μεγάλης ε, σημασίας για την Κεντρική Αμερική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία έχουμε την ίδια την πολιτική βαρύτητα αυτή τη συμφωνία, γιατί πρόκειται για μια πρώτη συμφωνία σύνδεση μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα και είναι σημαντικό βήμα συνεργασία με τι περιοχέ αυτέ. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια συνάντηση η οποία θέλει να, τονίσει την, να ενισχύσει την εμπορική ανάκαμψη της ε, Κεντρικής Αμερικής. Επίσης, ε, όσον αφορά το Παναμά, αφορά επίση την κοινωνική ένταξη, γιατί υπάρχει ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όλα αυτά δείχνουν την σταθερή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσει τις περιοχές αυτές. Όσον αφορά την εμπορική ολοκλήρωση, η συμφωνία θα προωθήσει τις επενδύσεις και θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο νομικής ασφάλειας που απουσιάζει τις συμφωνίες μεταξύ ορισμένες χώρες, αλλά είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Στην περίπτωση αυτή των δύο περιοχών, Υπάρχουν πολιτιστικές σχέσεις που θέλουμε να ενισχύσουμε για να υπάρξει μια ανταλλαγή υπηρεσιών που θα μπορέσει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση. Δεν θα ήθελα να παραλείψω να τονίσω μια σημαντική πτυχή της συμφωνίας που θα προωθήσει τις εμπορικές ροές και θα ενισχύσει τις επενδύσεις, τις διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και γεωγραφικών ενδείξεων σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Επίσης, οι φυτογεωνομικοί κανόνες του ΠΟΕ υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας. Η... Όλα αυτά μέτρα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την κοινωνική συνοχή όσον αφορά ε, την ρήτρα διασφάλιση και το μηχανισμό σταθεροποίηση για τι ε, μπανάνε. Μεταξύ των τροπολογιών έχουν συμπεριληφθεί ορισμένε τροποποιήσει που θεωρούσαμε ότι είναι ενδεδειγμένε για να βελτιωθεί αυτή η συμφωνία. Πράγματι, όπως είπα, σε σχέση με την ρήτρα διασφάλισης και το μηχανισμό σταθεροποίησης για τις μπανάνες, ε, είπα ήδη ότι οι τροπολογίες, τις τροπολογίες που εκείνες τροποποιήσεις που θεωρήσαμε ότι είναι ενδεδειγμένες για να βελτιωθούν αυτές οι τροπολογίες. Με αυτές και θεωρούμε ότι θα πρέπει να... Με τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η μελέτη και η εφαρμογή ε, του έργου του εποπτικού έργου τη Κομισιόν. Από την άλλη, ανταγωνικά τη σημασία που έχει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναπτύξει κάποιου προβληματισμού για τι επιπτώσει που θα έχει η συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζοντα ότι ο Οργανισμό δεν είναι ο καλύτερο δυνατό τόπο για να συμπεριληφθούν όλε μα οι ανησυχίε, θα θέλαμε παρόλα αυτά να τι λάβει υπόψη της η Επιτροπή. Τέλο, και επωφελούμενη από την παρουσία τη Επιτροπή στην αίθουσα, θα ήθελα να τη δείσω να μα πει πώς εκτιμά ότι θα εξελιχθεί η διαδικασία αυτή πέραν του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Ο κύριος Λάχτφριτ ε, ήταν ο εισηγητής, αλλά θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Ο Γιώργ Λάχιτφριντ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί γιατί έχει μια σημαντική συνάντηση στην Αυστρία και γι' αυτό με παρακάλεσε να τονίσω τα σημαντικά σημεία όσον αφορά τις αλλαγές ε, σε σχέση με τη διμερή ρήτρα διασφάλισης ε, και μηχανισμού σταθεροποίησης για την Κεντρική Αμερική. Έχουν κατατεθεί άλλες 16 τροπολογίες που χονδρικά ευθυγραμμίζονται με την γραμμή του εισηγητού και υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες όπου θα πρέπει να γίνει ένας λεπτομερέστερος έλεγχος κατά πόσο οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ε, υπερβαίνονται. Και υπάρχουν ε, ορισμένοι τομείς αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής και του Συμβουλίου που ε, θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Στόχος θα πρέπει να είναι να υπάρξει μία ε, ρήτρα διασφάλισης και ένας μηχανισμός σταθεροποίησης σε συμφωνία με την πολιτική μας. Τώρα, οι τροπολογίες ε, που υποβλήθηκαν για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις ε, πτυχές της βιωσιμότητας θα πρέπει να διαφυλαχθούν οπωσδήποτε και ή δυνατόν ε, και με την επιφύλαξη του νομικού τους ελέγχου να παραμείνουν. Η εξέταση των τροπολογιών, ιδιαιτέρως ε, από την νομική υπηρεσία και άλλους νομικούς ειδικού, θα ολοκληρωθεί πιστεύω σύντομα και με τον τρόπο αυτό θα διευκρινιστούν οι ε, τα κρεμόντα ερωτήματα και στη συνέχεια ο κύριος Λάιχτφριτ θα προτείνει κάποιους συμβιβασμούς ούτε ώστε δυνατόν να μπορέσουμε από κοινού να βρούμε μια διατύπωση των ε, προθέσεων των ε, συναδέλφων. Ε, συνολικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ καλή συνεργασία και υποθέτω ότι τελικά θα μπορέσουμε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση και για τα δύο θέματα. Η θέση μας όσον αφορά την ίδια την εμπορική συμφωνία και κανονισμός επίσης σχέση με την ρήτρα διασφάλισης δεύτερον. συνάδελφος Μακαλάρκιν από την ομάδα ΕΣΥΑΡ έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Συμφωνία Σύνδεσης είναι μια καλή συμφωνία και για τις δύο πλευρές. Το άνοιγμα στις υπηρεσίες, στους διαγωνισμούς, στις επενδύσεις υπερβαίνει και τη συμφωνία στις ε, εμπορικές σχέσεις και το πλαίσιο του ΠΟΕ θα μπορέσει έτσι να υπάρξει ένας ε, καλός διάλογος ε, στο πλαίσιο αυτό και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και σε θέματα όπως είναι κατά πολέμηση των ναρκωτικών, ε, η ασφάλεια κτλ. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επωφεληθεί, αλλά είναι αμφίδρομη η σχέση, γιατί θα έχουμε και εμείς πρόσβαση σε 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Ξέρουμε από μια ανεξάρτητη μελέτη αντικτύπου και βιωσιμότητας ε, με την αύξηση κατά 2,6 δι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση θέσεων εργασία, ευημερία, μείωση τη στόχιας και αυτό είναι ένα ακόμη λόγο να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία σύνδεσης. Όμως το σχέδιο έκθεσης για την υλοποίηση της ε, ρήτρα διασφάλισης μηχανισμού σταθερότητα τη μπανάνες μπορεί να στηριχθεί σε δρες γραμμές. Με ανησυχεί όμως ε, ο προστατευτισμός που επιδιώκεται για κάποιες ε, άκρως περιφέρειες της Ένωσης. Δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν προς όφελος ε, της συμφωνίας να παραταθεί μετά τον Ιανουάριο του 2020 ο μηχανισμός σταθεροποίησης που δεν προοριζόταν να είναι μόνιμος μηχανισμός και ίσως αυτό θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη την συμφωνία. Ούτε με ικανοποιεί ιδιαίτερα αυτό που λέγεται για τη σοβαρή είναι Παράγραφος Ένα, γιατί θα μπορούσε ή τόσο φαίνεται να υπονοείται ότι για να υλοποιηθεί ο μηχανισμό θεραπεία, να μην είναι τόσο αυστηρά τα κριτήρια, λέει πολύ σοβαρή βλά, very serious injury. εν κατακλείδη στηρίζω τη συμφωνία σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής και ελπίζω να υπογραφεί προς όφελος ε, και των ε, δύο πλευρών. Απλά φοβάμαι λίγο τις ε, επιπτώσεις που θα είχε ένας μεγαλύτερος προστατευτισμός, γιατί αυτό θα είχε ένα αποτέλεσμα για όλη τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να μιλήσω για τη ρήτρα διασφάλισης. Καταθέσαμε μια τροπολογία ακριβώς ε, με τα για τα κριτήρια αυτά, ε, τα προστατευτικά, για τα οποία είπε και η προϊολαλή σας, ε, για τις άκρους αποκέντρες περιφέρειες που θα πληγούν. Ε, με αυτή τη ρήτρα διασφάλιση που προτείνω σε αυτή την τροπολογία, ε, μάλλον λέμε ότι θα έχει ω στόχο να δημιουργηθεί ένα αυτόματο μηχανισμό για διαβουλεύσει. Σε αυτέ οι από περιφέρειε περιφέρειες ε, ουσιαστικά ζουν από αυτή την παραγωγή και μόνο. Η ρήτρα διασφάλιση η οποία εγκρίθηκε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα προϊόντα μας, αυτό που θα πρέπει να έχει ω στόχο είναι να ξεκινήσει άμεσα ε, τη διαδικασία διαβούλευσης, γιατί αυτές, επαναλαμβάνω, οι περιφέρειες πλήττονται. Και όταν ξεκινήσει η συζήτηση αυτή, ο διάλογος ε, και δεν ε, λαμβάνονται μέτρα προστασίας. Νομίζω ότι το άρθρο 12, σημείο 4 της τρίτας διασφάλισης πρέπει να εφαρμοστεί. Επίσης, νομίζω ότι θα ήταν αυτό πιο συνεπέζει με την εφαρμογή της ρήτρα, όπως αυτή εγκρίθηκε στο κοινοβούλιο μας. Now, ε, συμφωνεί με την Κόρεα. Υπάρχουν ε, άλλοι συνάδελφοι. Όχι. Άρα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γκάσπαρ Φροντίνη. Πού είστε? Είστε ο Κάσπαρ Φροντίνη ή όχι τελικά. Ε, κοιτάξτε, επειδή οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούν τη διασφάλιση, να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου που είναι πιο αρμόδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Wolfgang Müller λέγομαι. Είναι η τελευταία φορά που θα λάβω το λόγο και εγώ και ο συνάδελφος Τζον ε, Κλάικ από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Γεωργία. Ο Τζον ε, θα σας μιλήσει για το μηχανισμό θεραπείας της μπανάνης και για κάποια άλλα θέματα. Ξεκινώ λοιπόν. Ο κύριος Λάγκε θύμισε τη σημασία του μηχανισμού διασφάλισης και τροπολογίες συμφωνούν με την FTA, τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Και όλο το έργο που έχει γίνει εδώ, οι τροπολογίες ε, είναι θετικές και πράγματι ε, αναλογίες υπάρχουν και με το κρεατικό μοντέλο της ρήτρες διασφάλισης. Ε, κάποιες φορές όμως ο διάβολος κρύβεται σε λεπτομέρειες και γι' αυτό θα ήθελα να σχολιάσω κάποια σημεία. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τις τροπολογίες για την Κεντρική Αμερική. Τρεις ομάδες ε, μπορώ να διακρίνω. Η μία ομάδα βλέπουμε ότι θέτει κάποιο βάρος ε, στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στην Κομισιόν. Μια άλλη ομάδα τροπολογιών λέει ότι χρειάζεται περαιτέρω έργο για να επιτευχθούν πλήρω οι στόχοι των τροπολογιών και τρίτη ομάδα. Πρόβλημα συμβατότητας με την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Ο Τζον θα ασχοληθεί με το τρίτο, ε, με την τρίτη θέση των τροπολογιών και εγώ θα ασχολήσω τις δύο πρώτες. Είπα ότι βλέπουμε λοιπόν να τίθεται ένα βάρο στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και στην Κομισιόν από την πρώτη εβδομάδα τροπολογιών. Στι τροπολογίε αυτέ βλέπουμε προτάσει για επιπλέον εκθέσει που θα πρέπει να στέλνει το κοινοβου... το... η Κομισιόν στο Κοινοβούλιο. Σίγουρα είναι σημαντικό εργαλείο για το Κοινοβουλίο εκθέσει, γιατί έτσι μπορεί να παρακολουθεί την υλοποίηση τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλάγων. Ταυτόχρονα, έκθεση όμω σημαίνει επιπλέον βάρο επιπλέον φόρτο για τη διοίκηση ε, σε μια περίοδο που κόβουμε, περικόπτουμε τους σπόρους. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λεπτή ισορροπία για να μπορέσουμε να συμφιλιώσουμε τους δύο αυτούς αντικρουόμενους ε, μεταξύ τους στόχους. Έχουμε λοιπόν έκθεση για την παρακολούθηση των απαιτήσεων, τροπολογίες 33 και 41. Εγώ θα σας αναφέρω παράδειγμα την τροπολογία 33 που θα πρέπει σύμφωνα με αυτήν να, αναφέρει η Κομισιόν για μια αξιολόγηση για τον αντίκτυπο ε, στην απασχολησιμότητα, στη μέση των προϊόντων, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές επιχείρησεις κτλ. κτλ. Και στους μικρούς παραγωγούς. Αυτό του είδους οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες στην Κομισιόν αντίθετα με τα στατιστικά στοιχεία της αγωγή, για παράδειγμα. Για να εκπονήσουμε λοιπόν μια τέτοια έκθεση, θα έπρεπε να στραφούμε σε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ε, να του ε, θέσουμε αυτές τις ερωτήσεις. Άρα θα πρέπει πραγματικά να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, αν θέλουμε να επιβάλλουμε ένα τέτοιο φόρτο και σε εμά αλλά και στους οικονομικούς παράγοντες. Δεύτερη δέσμη τροπολογιών. Εκεί βλέπουμε ότι ίσως να χρειαστεί περισσότερο, ε, περισσότερες εργασίες να χρειαστεί, για να αντιμετωπίσουμε τα αιτήματα αυτών των τροπολογιών. 32 τροπολογία, 36, 40. Θα σας αναφέρω ως παράδειγμα την τροπολογία 36. Ο στόχος της τροπολογίας 36 είναι να οριστεί η έννοια σοβαρή επιδείνωση στι πιο απόμακρε περιφέρειε. Καλό είναι αυτό γιατί έτσι έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Σοβαρή επιδείνωση, serious deterioration, είναι μια προϋπόθεση για την επιβολή μέτρων διασφάλισης, τα οποία θα περιορίζονται σε συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχει και έννοια όμως serious injury, σοβαρή βλάβη. Αυτή είναι έννοια ενός κατοφλίου για να εφαρμοστούν μέτρα σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Αυτή η έννοια είναι πολύ απαιτητική. Μπορούμε να την πετύχουμε, αλλά είναι πιο απαιτητική σε σχέση με την άλλη έννοια του serious deterioration, Σοβαρή επιδείνωση. Αν βάλουμε τώρα την έννοια serious injury, σοβαρή βλάβη, ή αν αναμίξουμε τις δύο έννοιες, ουσιαστικά δυσχεραίνουμε την επιβολή μέτρων για μια πρόκεντρη περιοχή, άρα ουσιαστικά δεν επιτυχάνουμε το στόχο μας. Θα ήταν καλό να υπάρξει μια περίοδος προβληματισμού λοιπόν πάνω σε αυτό. Επίσης, τροπολογής 38 και 39 προτείνεται σε αυτές το Κοινοβούλιο να μπορεί να έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ε, δρομολόγηση μιας έρευνας. Ε, θα σας πω τι κάναμε στην περίπτωση της Κορέας. Ε, είναι καλό να δούμε το παράδειγμα της Κορέας και ενδεχομένω να ακολουθήσουμε την ίδια λύση. Ο Τζον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η πρόθεση του Κοινοβουλίου δεν θα είναι να υποβάλει τροπολογίες που θα είναι σε σύγκρουση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε σχέση επίσης με την τήρηση μιας θεμελιώδης ισορροπίας. Και υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, πολλές ε, προταθήσεις τροπολογίες που, θα είναι, που δεν είναι συμβατές ε, με την ουσία της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Και το πρώτο βήμα ε, είναι το εξής. Οι τροπολογίες που έχουν προταθεί για να υπάρξει μια διεύρυνση πέραν του 2020 ε, όσον αφορά το μηχανισμό σταθεροποίησης της μπανάνας. Είναι οι 34, 35 και 36. Ο μηχανισμός σταθεροποίησης ε, προτίθεται να είναι μια προσωρινή διάταξη για αυτή τη μεταβατική περίοδο της ε, μείωσης των ε, δασμών και να μην έχει μόνιμο χαρακτήρα. Και νομίζω ότι οι εταίροι μας της Κεντρικής Αμερικής δεν θα συμφωνούσαν ούτε καν σε δυνατότητα να γίνει μόνιμος αυτός ο, ο μηχανισμός. Βεβαίως, μετά το 2020 μπορούν να προστρέξουν στο γενικότερο μηχανισμό. Τώρα, όσον Υπάρχουν κάποιες άλλες τροπολογίες που είναι επίσης σύγκρουση με τις φιεστικές ε, δεσμεύσεις της ε, πολιτικής για την ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Οι τροπολογίες που προτείνουν να εφαρμοστεί αυτόματα η ρήτρα διαφύλαξη για τις μπανάνες αυτή τη στιγμή ε, έχουν επιτευθεί ορισμένα ορισμένοι όγκοι εμπορίου. Είναι οι τροπολογίες 34 και 33 που δημιουργούν σημαντικά νομικά προβλήματα. Δηλαδή, οι εταίροι μας στην Κεντρική Αμερική καταρχήν δεν έχουν συμφωνήσει ότι ο μηχανισμός σταθεροποίησης μπανάνας θα εφαρμοστεί αυτόματα αυτή τη στιγμή έχουν επιτευχθεί αυτά τα νότατα επίπεδα και δεν θα υπάρξει επραγμάτευση με τους εταίρους μας. Ε, τώρα, όσον αφορά την αυτόματη εφαρμογή του μηχανισμού σταθεροποίησης της μπανάνας θα τον μετέτρεπε ε, σαν ένα μηχανισμό ποσοστώσεων επί των εξαγωγών και δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στην επιβολή ποσοστώσεων όσον αφορά τις εξαγωγές μπανάνας. Άρα υπάρχει εδώ μια έλλειψη συμβατότητας. Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζουμε πλήρως πόσο ευαίσθητος είναι ο τομέας αυτός για ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς λόγω αυτού του ευαίσθητου χαρακτήρα η συμφωνία δεν απελευθερώνει πλήρως το εμπόριο της μπανάνας. Θα υπάρξουν ε, δασμοί, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεύτερον, θα διαπραγματευτούμε αυτό τον ειδικό μηχανισμό ακριβώς για τις μπανάνες, μόνο για τις μπανάνες. Και δεύτερον, όπως είπε ο Βόλφκαν, έχουμε προβλέξει ορισμένε ε, διατάξεις οι οποίες είναι προσαρμοσμένες σε εξόχως απόκεντρες ε, περιοχές της Ευρώπης Άρα πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσονται όλες οι ευαισθησίες ε, στις διατάξεις αυτής της συμφωνίας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα επανέλθουμε στους ε, εισηγητές Η Μαρία Κορέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη για να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τη συμβολή τους σε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη μεγάλη σημασία που έχει αυτή η Συμφωνία για την Κεντρική Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ε, κύριε Λάγκε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Και εγώ ήδη είπα ότι υπάρχουν θέματα όσον αφορά τη συνέπεια με των τροπολογιών μας και το νομικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να γίνει σχετικός έλεγχος. Παρ' όλα αυτά ε, θεωρούμε ε, ότι εκεί που υπάρχει νομιμότητα θα ε, μείνουμε στις τροπολογίες μας και ο κύριος Λάιχτφριτ πρόκειται να υποβάλει και περαιτέρω τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Τώρα στο χρονοδιάγραμμά μας έχουμε ήδη λάβει μια σχετική απόφαση για τον κανονισμό και την γνωμοδότηση για την ίδια τη συμφωνία και θα ήθελα να σας ενημεράσω ότι η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι η, αποφάση, η σχετικά με το σύνολο της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης θα ληφθεί από την ΑΦΕΤ. Άρα λοιπόν μας στερεί την αρμοδιότητα να λάβουμε εμείς μια απόφαση για αυτές τις εμπορικές συμφωνίες, κάτι που κατά την άποψή μου είναι παράδεκτο. Παρ' όλα αυτά, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι η ΑΦΕΤ θα πρέπει να ξεκινήσει μια έκθεση πρωτοβουλίας πριν από αυτή τη ε, διαδικασία λήψης απόφασης και εμείς ως συνδεδεμένη επιτροπή βάσει του ε, σχετικού άρθρου ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με την ΑΦΕΤ. Ε, δεν ξέρουμε πότε θα ληφθεί η σχετική απόφαση της ΑΦΕΤ και κατά πόσο θα συμμορφωθούν με την απόφαση αυτή της διάσκεψης των Προέδρων. Γι' αυτό λοιπόν ας αναμένουμε την ε, σχετική απόφαση. Εμείς ε, θα συμμετάσχουμε ως συνδεδεμένη επιτροπή. Ωραία, λοιπόν, και θα καταρτιστεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Τώρα, άρθρο, ε, ε σημείο υπαριθμών 8 της ημερήσιας διάταξης. Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κολομβίας και Περού. Δεν πρόκειται εδώ για μια συμφωνία σύνδεσης, άρα δεν θα αμφισβητηθεί η δική μας αρμοδιότητα εκ μέρους της ΑΦΕΤ στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν, εμείς είμαστε αρμόδια επιτροπή για το μηχανισμό σταθεροποίησης και τη ρήτρα διασφάλισης με την οποία θα ξεκινήσουμε. Ο Μάριο Νταβίτ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ε, δυστυχώς σε 20 λεπτά θα πρέπει να φύγω. Εάν μπορούμε να αλλάξουμε την σειρά, παρακαλώ, της συζήτηση. Θα σήμουν ευγνώμων. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι. Ας αλλάξουμε λοιπόν το άρθρο 8 και 9 που αφορά την ίδια τη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Κολομβίας και του Περού εφετέρου ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Μάριο Νταβίτ από το ΕΛΚ. Πρόκειται για μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. στο Συμβούλιο των Υπουργών δεν έχω ακόμα την πολιτική έγκριση για αυτή τη συμφωνία και αναμένουμε την επίσημη απόφαση. Και αυτό θα γίνει περίπου στα τέλη Μαΐου. Παρόλα αυτά, εμείς ε, είχαμε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και αυτή είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Μάριο Νταβίτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι αποφασίσαμε να αποδεχθούμε την πρόταση των σοσιαλιστών και δημοκρατών να υποβληθεί μια προφορική ερώτηση συμβασμού προς την Επιτροπή που πιστεύουμε ότι είναι σημαντική και παρουσιάστηκε από την Ίντα και θα ε, εγκριθεί αύριο, ελπίζω, το προφορικό αυτό ερώτημα εδώ στην Επιτροπή. Και ελπίζουμε ότι θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα της δεύτερης ολομέλειας του Μαΐου του Στρασβούργου. Θα πρέπει να υπάρξει μια πρόταση ψηφίσματος για να συμπεριληφθούν εκ των προτέρων, δηλαδή πριν από τη συγκατάθεσή μα το Σεπτέμβριο, οι κοινέ θέσει όσον αφορά τι εμπορικέ και μη εμπορικέ ε, πτυχέ. Ένα πρώτο σχέδιο αυτού του ψηφίσματο θα κυκλοφορήσει σύντομα, πιστεύω στι αρχέ τη προσεχού εβδομάδα και στη συνέχεια μπορούμε να ορίσουμε την ημερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών, κύριε Πρόεδρε οι υπηρεσίε μου είπαν ότι, οι υπηρεσίες μου είπαν ότι θα πρέπει να κατατεθούν οι τροπολογίες για να μέχρι τέλη Μαΐου το μεσημέρι για να μπορούν να μεταφραστούν. Επίσης ψηφίσαμε, θα ψηφίσουμε ένα ψήφισμα ε, το Μάιο με την ΙΝΤΑ, ούτως ώστε να μπορέσει να εγκριθεί το κείμενο πριν από την τελική ψηφοφορία του κειμένου τον Ιούνιο στο Στρασβούργο. Καταβάλουμε μια προσπάθεια, κύριε Πρόεδρε, ε, και προσπαθούμε να έχουμε όλες τις εισφορές και κοιτάω το David Martin, όλες εννοώ, ούτως ώστε να έχουμε μια πραγματική προοπτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την συμφωνία που θέλουμε να είναι υποδειγματική με τις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες, τις οποίες θέλουμε να θεωρούμε ως εταίρους και όχι απλούς αποδέκτες των δικών μας θέσεων ή επιταγών. Ε, νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να πατρονάρει αυτές τις χώρες που εκουσίως αποφάσισαν να είναι οι δικοί μας εταίροι. Οι εταίροι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν το ισότιμα. Δυστυχώς ακούω ορισμένε φορές μερικές παρεμβάσεις που φαίνεται οι ομιλητές να γνωρίζουν περισσότερα για τις χώρες αυτές από τους κατοίκους αυτής της χώρας. Επίσης άκουσα κάποια αιτήματα από συναδέλφους να επιβάλλουμε στις τρίτες χώρες ε, πράγματα τα οποία δεν επιβάλλουμε καν στις δικές μας χώρες και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό γελιοποιούμεθα. Για δείτε τι γίνεται με τη σύμβαση 1.6 ε, που δεν έχει υπογραφεί, ε, τη σύμβαση ILO, συγγνώμη, η οποία 1.8.5 ε, η οποία ακόμα δεν έχει υπογραφεί από τρεις χώρες μέλη και αφορά τα, τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα συλλογικής ε, διαπραγμάτευσης. Αυτό μου θυμίζει την κατάσταση πριν από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Και ε, πιστεύω ότι θέλουμε να είμαστε θετικοί και να έχουμε σεβασμό προς όλους μας τους ε, εταίρους, λειτουργώντας αξιόπιστα, καλόπιστα. Τώρα, όσον αφορά τις ίδιες τις συμφωνίες, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για το ψήφισμα. Η Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ Κολομβίας και Ηνωμένων Πολιτειών θα τεθεί σε ισχύ στις 15 Μαΐου ήδη, δηλαδή σε μερικές εβδομάδες. Θα ήθελα να σας το επενθυμίσω. Και θα ήθελα να σας πω ότι τόσο η Κολομβία όσο και το Περού κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για να βελτιώσουν τις γενικές συνθήκες των πολιτών τους, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα και βιώσιμη ανάπτυξη και ευτυχώς παρά όλες τις ε, ε, σοβαρές ε, προσπάθειες εκ μέρους των πολιτών, της κυβέρνησης, των οργανισμών, των μη κυβερνητικών οργανισμών. Ε, δυστυχώς θα πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά ακόμα και στην Κολομβία και στο Περού όσον αφορά την κατάρτιση του νέου νομοθετικού πλαισίου το οποίο προτίθεται να επιλύσει όλα τα μακρά προβλήματα που έχουν σαν συνέπεια τη φτώχεια, τη διαφθορά, τον ε, εμφύλιο, τις ε, σειράξεις με ένοπλες ομάδες, ε, ε των ενόχων για εγκλήματα κλπ. Είναι γεγονός ότι τόσο η Κολομβία και το Περού παρόλα αυτά έχουν κάνει σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια και αφού ο, κύριος, ο Ντεσάντς έγινε κύριος, ο, ο καινούριο πρόεδρος και θα ήθελα να σας παραθέσω τα όσα είπε η Amnesty International στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών που έλαβε χώρα στη Γενέβη τον περασμένο μήνα. Είπε τα εξή. Ε, ε, η, κυβέρνηση της Κολομβίας θέλει να θέσει ένα τέλος ε, στην ατιμορρησία η σχέση της κυβέρνησης με τους οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, γενικά υπήρξε οικοδοματική, ιδιαίτερος ε, εάν τη συγκρίνουμε με, τις προηγούμενες, με την εργασία των προηγούμενων κυβερνήσεων. Επίσης, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει κάποιες πολιτικές υπέρ των θυμάτων των ένοπλων σειράξεων και ε, ιδιαίτερα στα δικαιώματα γης εφόσον εφαρμοστούν σωστά θα είναι ιδιαίτερως ευεργετικά για τους κατοίκους της χώρας, ούτως όταν τους επιστραφούν ε, οι περιοχές ε, ε, που τους έχουν αφαιρεθεί παράνομα. Θα πρέπει να λάβουμε γνώση ότι τα τελευταία χρόνια στην Κολομβία υπάρχουν πάρα πολλές δολοφονίες συνδικαλιστών. Ε, το 2011 ήταν 26 περιπτώσεις ε, δολοφονίας. Παρόλα αυτά υπάρχει δηλαδή μια σημαντική μείωση, την περασμένη χρονιά ήταν 50 τόσες. Υπάρχει μια σημαντική μείωση, παρόλα αυτά είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός των δολοφονιών. Η Κολομβία, όπως σας είπα, έχει εφετήσει ε, μέτρα για να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα και υπάρχει μεγάλος αριθμός αύξησης αρμόδιων ανακριτών και εισαγγελέων για εγκλήματα που απευθύνονται ειδικά σε συνδικαλιστές. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αύξηση του αριθμού αυτών των ανθρώπων. Η καταπολέμηση της ατιμορρησίας είναι επίσης ένας από τους μείζονες στόχους αυτής της κυβέρνησης και σύμφωνα με την ILO μεταξύ του 10 και του 11 υπήρξαν 28 ε, καταδίκες και περίπου 400 πολίτες ε, καταδικάστηκαν για τέτοιου είδους εγκλήματα. Άλλο σημαντικό μέρος, ε, μέτρο είναι ένα πρόγραμμα προστασίας το οποίο εξασφαλίζει προστασία σε πάνω από 11.000 πολίτες εκ των οποίων πολλοί είναι συνδικαλιστές, 11% είναι δημοτικοί σύμβουλοι 18% είναι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 4% είναι δημοσιογράφοι. Και το πρόγραμμα αυτό ε, το 11 έχει ένα προπολογισμό 220 εκατομμυρίων. Τέταρτον, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της διατήρησης του επικοδομητικού διαλόγου με, τις, ε, με τους εταίρους μας όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των προδιαγραφών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και γι' αυτό καλωσορίζω την έναρξη του αμοιβαίου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που άρχισε το 2009 μεταξύ Κολομβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συναντήσεις που γίνονται δύο φορές το χρόνο και είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας είναι ανοιχτή για το διάλογο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς ε, και με άλλες χώρες. Επίσης, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός είναι ότι η συμφωνία περιλαμβάνει δεσμευτικές και περιεκτικές διατάξεις όσον αφορά τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αναφέρεται στο άρθρο 1, παρθέτω σχετικό απόσπασμα, επελαμβάνει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι όπως κατοχυρώνονται στην ε, Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, στην, ε, ένομη, και στο κράτος, του κράτους δικαίου. Ο σεβασμός αυτών των δικαιωμάτων συνιστά θεμελιώδες στοιχείο της συμφωνίας. Ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστά κατάφορη παραβίαση της ε, συμφωνίας ε, εμπορίου και θα μπορούσε να οδηγεί στη λήψη των αναγκαίων μέτρων συμπεριλαμβανόμενης και της δυνατότητας ε, μερικής ή πλήρους αναστολής της εμπορικής συμφωνίας και αυτό είναι εξόχως ε, δεσμευτικό. Τέλος, η Συμφωνία Δέσμευσης παρέχει επαρκείς εγγύησεις ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συμφωνια Δέσμευση παρεχει επαρκεις εγγυησεις ουτως ωστε αρχιτεκτονική των εμπορικών αυτών σχέσεων κινείται προς την κατεύθυνση μιας αύξησης περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης προωθώντας και διαφυλάτοντας ένα υψηλό επίπεδο εργασίας και περιβαλλοντικού σεβασμού από όλες τις πλευρές και περιλαμβάνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά τι εξελίξει αυτέ, ε, θα θέλαμε να προτείνουμε μια ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στην παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γέννη, των εργασιακών δικαιωμάτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλε τι χώρε εταίρου μα. Επίση, προτείνουμε ε, υπό, σε σχέση με τις νέες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες να οργανωθεί μια δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και μετά από την ακρόαση αυτή να υπάρξει μια γραπτή έκθεση η οποία θα υποβληθεί στην Επιτροπή ΙΝΤΑ και στην Υποεπιτροπή σε σχέση με τα αποτελέσματα ε, εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών μέχρι τώρα. Τέλος, και με αυτό θα καταλήξω, πιστεύω ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε αυτή τη συμφωνία σαν ένα εργαλείο αλλαγής μέσω της προσέγγισης. Η πραγματικότητα αλλάζει στις μελλοντικές χώρες εταίρους μας, παρόλο που ορισμένοι μένουν να το παραγνωρίζουν. Μαζί με τη σχηνόμενη διαδικασία επικύρωσης θα ήθελα να πω ότι είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από τη στάση του Περού όσον αφορά με τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις και τις σωστές διαδικασίες που υιοθέτησε το Περού ε, σε σχέση με αυτό. Ο Επίτροπος είπε ότι έστω και αν η συμφωνία υπογραφεί από όλες τις χώρες μέλη, δεν υπάρχει η πρόθεση να μπει η τελική υπογραφή της Κομισιόν έως ότου επικυρωθεί ένας επαρκής αριθμός γεωγραφικών ενδείξεων, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Περού. Και εάν το λέω σωστά, έχουμε 160 ενδείξει που είναι κόκκινη γραμμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Κολομβία ήδη το έχει πράξει, αλλά οι περβεγενοί φίλοι μας είναι περίπου στο 50 και ε, σε σχέση με τις εμπορικές πτυχές της σύνδεσης δεν ε, ήταν να υπάρχει κανένα σχόλιο στην προηγούμενη σχετικό σχόλιο στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ελπίζω ότι μπορώ να έχω την ειλικρινή υποστήριξη για αυτό το ψήφισμα και επίσης για το σχέδιο πρόταση που θα ακολουθήσει όσον αφορά την ε, συγκατάθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ αναλυτική αυτή η παρουσίαση. The EU Colombian Peru trade Σε σχέση με αυτές τι συμφωνίες με το Περού και την Κολομβία. Προφορική ερώτηση Λάγκη και Μάριο Ντάβιτ. Την έχετε στο φακελό σας την ερώτηση αυτή. Και θα τη μελετήσουμε πριν ε, την υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο. Επόμενος είναι ο Μπερν Λάγκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πρόκειται για ένα ψήφισμα το οποίο συνδέεται με ένα ερώτημα στην Επιτροπή και ε, με το σκοπό να διευκρινιστούν κάποιες ασάφειες που παραμένουν και να εντοπιστούν κάποιες αδυναμίες της ε, συμφωνίας και πράγματι είμαστε πεπισμένοι ότι στην εμπορική συμφωνία υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι απολύτως ε, ξεκάθαρη η αρχή ότι το εμπόριο δεν είναι μια πολιτική αυτή καθ' αυτή, αλλά θα πρέπει να συμβάλλει ούτως ώστε να βελτιώνεται η κατάσταση των πολιτών στις ε, χώρες που διενεργούν εμπορικές συναλλαγές. Και υπό την έννοια αυτή θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια πράγματα και να δούμε σε ποιο βαθμό επιπρόσθετα προς τις εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να συνάψουμε κάποιες συμφωνίες που να ανταποκρίνονται σε αυτή την αρχή, δηλαδή ε, να εξυπηρετεί των, ε, τις δικές διαβίωσης των ανθρώπων Στι χώρε μεταξύ των οποίων συνάπτουν αυτέ τι συμφωνίε. Γι' αυτό το ζητούμενο είναι να σκεφτούμε ακριβώ σε ποιου τομεί επιθυμούμε μια, την επίτευξη μια επιπλέον συμφωνία. Και είναι απολύτω ξεκάθαρο ότι στην Κολομβία κινούνται τα πράγματα. Αυτό είναι πέραν πάσης αμφισβητήσεως και θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά και πιστεύω ιδιαίτερα ότι ο νόμος περί θυμάτων είναι ένα καθοριστικό βήμα για να επιτευχθεί η ρήνευση στην Κολομβία και με την, έναρξη, με την αρχή της εφαρμογής σε αυτό το έτος έχουν γίνει τα πρώτα βήματα ούτως ώστε να καταπολεμηθεί η εκδίωξη των ανθρώπων από τη γη τους και να τους επιστραφούν αυτές οι γέες. Αυτή είναι μια καλή ένδειξη για το ότι κινούνται τα πράγματα αυτά και πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία αλλαγή στην Κολομβία θα πρέπει να συνοδευτεί και να ενισχυθεί από επιπλέον ε, συμφωνίες. Αυτό θα πρέπει να είναι, αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μου. Και όταν ε, μιλώ για συμφωνίες, ε, θα ήθελα να το συνοδεύσω με τρεις προβληματισμούς. Αναφίβολα στην συμφωνία αναφέρεται ότι η Κολομβία, η Περού και, το Περού συγγνώμη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται στην ε, Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό λέει τα πάντα, αλλά ταυτόχρονα κύριοι συνάδελφοι απολύτως τίποτε, γιατί δεν εξεδικεύεται στη γενική αυτή αρχή ε, ε, ποιες είναι οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν εδώ. Και δεύτερον, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται κανένας απολύτως μηχανισμός ε, επίβλεψη παρακολούθησης. Ποιος επαγρυπνεί για την τήρηση αυτής της γενικής αρχής. Άρα λοιπόν έχω την πεποίθηση ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία παρακολούθησης όσον αφορά την τήρηση αυτών των γενικόλογων διατάξεων. Ε, και επίσης υπάρχει και το ερώτημα του τι θα γίνει αν το ένα μέρος, συμβαλόμενο μέρος διαπιστώσει, γιατί μπορεί η Κολομβία να διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται κάποιες διατάξεις στην Ευρώπη. Τι θα πρέπει λοιπόν ε, να συμβεί εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Και υπάρχει η δυνατότητα να ανασταλεί η συμφωνία, αλλά αυτό είναι δυνατόν να γίνει μόνο εφόσον υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο. Και με όλο το ρεαλιστικό πνεύμα που επιδεικνύουμε δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτή, αυτός είναι ένας επαρκής ε, χειρισμός, με επαρκή αντιμετώπιση αυτής της ε, διάταξης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα της ε, παρακολούθησης, της επίβλεψης, της επαγρύπνησης για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δεσπιστεί ο αντίστοιχος μηχανισμός και επίσης θα πρέπει να υπάρξει και ένα μηχανισμός διαθέτηση των διαφορών. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο αναφέρεται στο 267 και 268 ε, άρθρα που αφορούν την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε συμφωνήσει στο άρθρο 1 το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά στο κεφάλαιο βιωσιμότητα έχουμε κάποιε εργασιακές προδιαγραφέ και κάποιε περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ. Και, και αυτές ε, ε, θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικότερα και στα άρθρα τα οποία προανέφερα λέγεται ότι η εφαρμογή αυτού του κεφαλαίου περί βιωσιμότητας εξαρτάται από τους ε, πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, ενώ η χρήση αυτών των κονδυλίων δεν δημοσιοποιείται καν. Άρα, τι συμβαίνει. Ναι, μεν λέμε, κάνουμε μεγαλοσχήμονες εξαγγελίες, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να τις εφαρμόσουμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει στο κεφάλαιο περί βιωσιμότητας, να υπάρξει διαφάνεια εν σχέση με τους διαθέσιμους πόρους και να προβλέψουμε μια διαδικασία βάση της οποίας θα εξευρεθούν περαιτέρω κονδύλια για την εφαρμογή. Συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το ζήτημα των επιθεωρητών εργασίας. Εάν δεσμευόμαστε για την τήρηση των βασικών προδιαγραφών εργασίας που θέτει η ΑΕΛΟ, το ζήτημα δεν είναι απλώς να προσχωρήσουμε στις βασικές αρχές του Παγκοσμίου Γραφείου Εργασίας, αλλά ε, και κύριε συνάδελφε, ε, είπατε ότι δεν έχουν καν ε, υπογράψει τη σχετική συμφωνία όλες οι χώρες μέλη. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι η υπογραφή, αλλά η εφαρμογή. Για παράδειγμα, το θέμα των επιθεωρητών εργασίες οι οποίοι ελέγχουν στις επιχειρήσεις τι γίνεται ακριβώς εκεί. Και αυτό είναι ένα θέμα πόρων και πάλι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να εφαρμόζονται τα ε, συμφωνηθέντα. Και ο τρίτο, το τρίτο μου σημείο αφορά την κοινωνία των πολιτών και τη συμμετοχή της. Έχω την πεποίθηση ότι η αξίωση μέσω κάποιων ενεργειών να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων ε, θέτει σαν ε, προϋπόθεση να εξετάζεται και το έργο των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων, της, της κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Κορέας, εκεί υπάρχουν κάποιες ενώσεις πολιτών που ε, συνεργάζονται μεταξύ τους και θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιοι παραπλήσιοι μηχανισμοί όσον αφορά ε, και να θεσπιστούν ε, συνοδευτικά με τη σύναψη της συμφωνίας ανεξάρτητες οργανώσει κοινωνία των πολιτών, οι οποίε να συνοδεύουν και να στηρίζουν τη διαδικασία εφαρμογή αυτών των συμφωνιών, να μπορούν δηλαδή να παράσχουν συμβουλέ ή να δέχονται παράπονα, ούτως ώστε να συνοδεύουν υποστηρικτικά και να οργανώνουν αυτή τη διαδικασία ει όφελο των πολιτών μη κυβερνητικοί οργανισμοί, εργοδότες και συνδικάτα να συνοδεύουν από κοινού αυτή τη διαδικασία. Και θεωρώ ότι εάν μπορούμε να διατυπώσουμε αυτές τις τρεις, ε, τα τρία σημεία σε ένα μνημόνιο ή σε ένα σχέδιο δράσης, δηλαδή σε μια πρόσθετη συμφωνία, πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να προσλάβει εντελώς διαφορετική μορφή εμπορική συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ρητά τους δύο εισηγητές για τον ε, ιδιαίτερο λεπτομεριακό τρόπο που ανέπτυξαν την προβληματική της συμφωνίας καθώς ε, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώπιον της διαδικασίας ε, επικύρωσης των συμφωνιών. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά πώς οι δύο έννοιες κλειδί που ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι εδώ, ε, το monitoring, η παρακολούθηση και το implementation, η εφαρμογή ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και όσον αφορά την εφαρμογή θα πρέπει να δούμε ε, ακριβώς, τι ακριβώς πρέπει να εφαρμοστεί. Ελέγχεται από τον εισηγητή ότι ούτε καν η σύμβαση της ILO δεν έχει υπογραφεί. Νομίζω ότι δεν, θα πρέπει, δεν είναι δυνατόν να κρίνουμε άλλους εάν δεν είμαστε ήδη εντάξει. Και νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να δούμε με μεγάλη σοβαρότητα τι γίνεται σχέση με αυτό. Δεύτερον, και αυτό αφορά επίση την εφαρμογή, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται ακριβώς στην πράξη. Και εάν διαπιστώσουμε ότι ακόμα και οι διαδικασία ατιμορρησίας που υπάρχει, κατάσταση ατιμορρησίας που υπάρχει στην Κολομβία τελικά ε, δεν έχει ε, αλλάξει ή δεν έχουν εφαρμοστεί οι αλλαγές που έχουν εξαγγελθεί. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά τι γίνεται ακριβώς και με εγκλήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί στο παρελθόν. Έστω ε, και αν ε, ο αριθμός των ε, δολοφονηθέντων συνδικαλιστών έχει μειωθεί ε, και πράγματι υπάρχει μια αλλαγή εδώ, αλλά όπως είπε ο κύριος Ντάβιτ, ο αριθμός αυτός παραμένει μεγάλη, μεγάλος. Πώς λοιπόν ε, ε, γίνεται η εφαρμογή. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και τα όσα είπε ο Μπέρντ ε, Λάγκε σε σχέση με την εφαρμογή των συμβάσεων δεν θα πρέπει να επιμείνουμε να γίνει αυτό πριν από την επικύρωση των εμπορικών συμφωνιών, ούτως ώστε να δείξουμε πιο καθαρά ότι μας ενδιαφέρει η κατάσταση των ανθρώπων στην ε, Κολομβία ή στο Περού, των ανθρώπων που ακριβώς ε, έχουμε σαν στόχο να αποφεληθούν από τις εμπορικές συμφωνίες. Τώρα, όσον αφορά το κεφάλαιο για την ε, βιωσιμότητα, ε, το κεφάλαιο αυτό δεν έχει ένα πραγματικά δεσμευτικό χαρακτήρα υπό την ε, έννοια μιας διαθέτηση των διαφορών. Και σε αντίθεση με τα όσα είπε ο κύριος Ντεκούχτ σε αυτή την επιτροπή, απουσιάζουν ακριβώς εκείνοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί ή δομές ε, όταν ε, υπάρχει μία διαθέτηση των υφρών, υπάρχει μία, υπάρχουν διαφορετικές ε, ερμηνείες. Και στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να δράσουμε κατάλληλα. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει επίσης να αλλάξει πριν από την τελική κύρωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο όνομα της τη εισηγήτριας, ε, κυρία Κατρίν Μπέρκ, θα ήθελα να κάνω κάποιε σύντομε παρατηρήσει σε σχέση με αυτήν την έκθεση. Δυστυχώ, δεν μπόρεσα να την έκθεση ε, Ούτω ή άλλω, ε, τι περισσότερε σημαντικέ παρατηρήσει τι υπέβαλαν ήδη οι συνάδελφοι Λάγκη και Σόλτ. Πάντω, για μα είναι σημαντικό να έχουμε μια θέση της κυβέρνησης της Κολομβίας, πολύ συγκεκριμένη δέσμευση, ότι θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάσταση των συνδικαλιστών, ειδικά στην Κολομβία, ώστε να υπάρξει μια στέρεα βάση για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις πολιτικές αλλά και εμπορικές μας σχέσεις. Πιστεύω πως αυτή η θετική τάση που διαβλέπετε τον τελευταίο καιρό θα πρέπει να στριφθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο. Υποστηρίζουμε την πρόταση του εισηγητή να υποβάλουμε προφορική ερώτηση προηγουμένως, πριν μάλλον αποφασίσει το Κοινοβούλιο ε, για τη θέση του ένα σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα να παρουσιαστεί και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε ένα λογικό μια λογική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Πιστεύουμε πως αυτό το, θα θέλαμε μάλλον αυτό το πρόγραμμα δράσης να παρουσιαστεί και να αρχίσει να εφαρμόζεται πριν από την έναρξη ισχύω Τη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών και επίσης, και νομίζω και αυτό αναφέρθηκε και είναι το πιο σημαντικό, ε, το σχέδιο αυτό να συμπεριλαμβάνει δεσμευτικές διατάξεις ε, ε, που να, όρους μάλλον δεσμευτικούς που να μπορούν να, να εξεταστούν και να αξιολογηθούν με αντικειμενικό τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ακούσουμε την Κομισιόν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να σχολιάσω κάποια από τα πράγματα και τα σχόλια που έγιναν. Καταρχήν, η Κομισιόν συμφωνεί πλήρως με την αξιολόγηση. Ξέρω ότι αναγνωρίζεται η πρόοδος που καταβάλει η Κολομβία στην δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση στην Κολομβία εδώ και πολλά χρόνια και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό, τα έχουμε ήδη πει. Τώρα η κυβέρνηση της Κολομβίας ε, θέλει να βελτιώσει την κατάσταση και έχει δεσμευθεί με τη, απέναντι στη διεθνή κοινότητα και απέναντι σε εμά για τη βελτίωση της κατάστασης. Ε, σε αυτό το πλαίσιο ε, βλέπουμε ότι η συμφωνία αυτή δίνει στην κολομβιανή κυβέρνηση και σε εμά ένα επιπλέον εργαλείο για να προχωρήσουμε σε αυτόν τον αγώνα ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία. Νομίζω λοιπόν πως μέσα σε αυτή την προοπτική θα πρέπει να δούμε την συμφωνία τούτη. Έχοντας όλα αυτά υπόψη και θα σας δώσω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, ε, καταρχήν ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις σχετικές ρήτρε, καθώς και τη δυνατότητα αναστολής της συμφωνίας εάν αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά η ρήτρα έχει συνταχθεί με ιδιαίτερα ευρύ τρόπο ώστε να δίνεται μέγα περιθώριο για ερμηνεία και να μην ε, και δεν προβλέπεται συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης για την εφαρμογή. Αλλά αυτή είναι η γραμμή που ακολουθείται για όλες αυτές τις συμφωνίες. Δεν θέλουμε να έχουμε μηχανισμούς που να περιορίζουν τις δυνατότητες ακτίμησης, αξιολόγησης για το τι είναι παραβίαση ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διατηρήσει το δικαίωμά τη να μπορεί να ενεργήσει, όποτε φαίνεται ότι υπάρχει παραβίαση, χωρί όμω να δεσμεύεται ή να περιορίζεται, να υποχρεώνεται από κάποιο συγκεκριμένο μηχανισμό ε, για το συγκεκριμένο αυτό τμήμα που είναι φυσικά πολύ ευαίσθητο από πολιτική άποψη. Δεύτερον, <clears throat> όταν μιλάμε για το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ακούστηκε ότι οι διατάξεις αυτού του κεφαλαίου δεν είναι δεσμευτικές. Όχι. Οι δεσμεύσεις αυτές είναι πλήρως ε, νομικά δεσμευτικές για την Κολομβία και για το Περού. Και σε αυτά τα κεφάλαια Κολομβία και Περού δεσμεύονται να εφαρμόσουν τα όσα συμπεριλαμβάνονται εκεί. Δεσμεύονται να εφαρμόσουν ε, τις ε, θεμελιώδεις συμβάσεις για περιεργασίας, περι, περιβάλλοντος να εφαρμόσουν τη δική τους νομοθεσία. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Είναι δεσμευτικές αλλά είναι ε, δυνατόν να επιβληθούν. Μάλιστα. Δεν ε, υπόκειται στη ε, μηχανισμό ρύθμισης διαφορών του συμφωνία, της συμφωνίας, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός διατησίας για το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Και αυτό γιατί διότι πιστεύουμε πως ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι πιο αποτελεσματικός ώστε πραγματικά να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να επιβάλλουμε την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων. Και γιατί αυτό, διότι όταν μιλάμε για τα εμπορικά θέματα, κανονικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο αντίκτυπος στο εμπόριο ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών για τα εμπορικά θέματα πρέπει να αποδεικνύει ότι υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο για το εμπόριο πριν μπορούμε να προβούμε σε δράση. Στο συγκεκριμένο τομέα είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι μια παραβίαση σε σχέση με κάποιες από τις δεσμεύσεις που έχουν για νομικές πτυχές ή για περιβαλλοντικές πτυχές έχουν όντως αντίκτυπο στο, στο εμπόριο. Και γι' αυτό η δυνατότητα να δράσουμε περιορίζεται. Έπειτα, για αυτού του είδους της δεσμεύσεις πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο πριν αρχίσουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις που είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποδείξουμε πως όντως υπάρχει εμπορικό στο εμπόριο λόγω της ε, ε, λόγω της παραβίασης να μπορούμε να έχουμε λοιπόν ε, ε, εκθέσεις από έναν ε, ανεξάρτητο εκτιμητή, στην, μια έκθεση στην οποία θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση του μέρους που κατηγορείται, να εξηγήσει πώς θα αντιμετωπίσει το, πώς θα χειριστεί το θέμα και ποια είναι τα βήματα που ε, στα οποία θα προβεί ώστε να εφαρμόσει οτιδήποτε περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Και όλα αυτά θα είναι ε, δημόσια. Νομίζουμε ότι στη συγκεκριμένη ε, περίπτωση είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ότι ο άλλος μηχανισμός που έχουμε για εμπορικά θέματα. Λοιπόν, είναι νομικός δεσμευτικό. Υπάρχει σαφής μηχανισμός επιβολής για αυτό το κεφάλαιο και πιστεύουμε πως αυτός ο μηχανισμός είναι προσαρμοσμένος στην ιδιαίτερη φύση των διατάξεων του συγκεκριμένου κεφαλαίου. So I, I think this, with this I cover uh, uh, most of the, of the Νομίζω πως έτσι τώρα έχω μιλήσει για τα περισσότερα θέματα που αφορούν την Κομισιόν ε, και βεβαίω για τις γραπτές ερωτήσεις θα τις περιμένουμε και θα απαντήσουμε σε αυτό το χρόνο. Λούση Αντρικένα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω και τους ε, δύο εισηγητές, Μάριο Ντέιβιντ και Λάγκε. Ε, θα ήθελα επίσης να πω ότι υποστηρίζω τη γραπτή ερώτηση στην ε, Κομισιόν για την ε, συμφωνία με την Κολομβία και το Περού. Κάποιες παρατηρήσεις για τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι τμήμα της συμφωνίας. Εγώ εργάζομαι από το 2005 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Λατινική Αμερική και ιδιαίτερα στην Κολομβία. Πολλές παραβιώσεις αναφέρονται και το θέμα αυτής τη εμπορική συμφωνίας πρόσφατα συζητήθηκε στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο εισηγητή Μάριο Νταβίντε ήταν παρόν και εκεί. Η Επιτροπή μας και ε, συγκεκριμένα εμείς ε, τονίσαμε τη σημασία της ύπαρξης ε, όρων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη όταν καθορίζει ρήτρε ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να είναι πλήρη και θα περιλαμβάνουν μηχανισμό ανάκλησης της συμφωνία σε περίπτωση που ο πολιτικός διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δυνατός. Γι' αυτό θέλω να καλωσορίσω το άρθρο 1 της συμφωνίας αυτής που ορίζει πως ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών του κράτους δικαίου όπως ορίζονται στην Παγκόσμια ε, Δήλωση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θα ισχύει. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση παραβιάζει τα συγκεκριμένα αυτά σημαντικά στοιχεία ή τα, τα, συμβαλόμενα μέρη θα μπορούν μονομερός και χωρίς ειδοποίηση να, ακυρώ, να στείλουν την ε, συμφωνία. Να τονίσω ότι αυτό το άρθρο στη συμφωνία δεν αρκεί, όπως αναφέρθηκε ε, και από άλλους συναδέλφους. Ο πολιτικός διάλογος όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, της δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου θα πρέπει να εξαντλώνται συστηματικά. Ε... Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε έναν διαρκή και ανοιχτό διάλογο με τις εν λόγω χώρες, να είμαστε δραστήριοι και να προβαίνουμε σε συγκεκριμένα βήματα στον αγώνα κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι δράσεις χρειάζονται όχι μόνο πριν από τη την υπογραφή της συμφωνίας, αλλά και για την, κατά τη διάρκεια της ισχύω αυτής της συμφωνίας και της εφαρμογής της, που πιστεύω πως θα επιφέρει ωφέλη και για τις δύο χώρες. Ναι, λοιπόν, υποστηρίζω αυτή τη συμφωνία, αλλά ταυτόχρονα θα περιμένω για την απάντηση της ε, ε, Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση. Και σε σχέση με τις, ε, την πρόταση κανονισμού. Α, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Διακόπτει ο Πρόεδρος, γιατί θα το εξετάσουμε μετά. Μάλιστα. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για την εμπορική συμφωνία. Ε, θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης 29 Μαΐου. Στοχεύουμε τον Ιούλιο για υιοθέτηση της έκθεσης αυτής στην Επιτροπή και το Σεπτέμβριο για την υιοθέτησή της στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ και τώρα πάμε πίσω στο σημείο 8. Εδώ έχουμε τον ε, κανονισμό ρήτρα διασφάλισης. Ε, ο εισηγητής είναι ο κύριος Λάγκεν. Έχω ένα πρόβλημα. Ο κύριος Ντάιβιντ είναι πολύ γοητευτικός. Ο κύριος όλοι το συμπαθούμε και εγώ μεταξύ όλων. Αλλά θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας αυτήν την άποψη. εφόσον είναι εισηγητής, καλό θα ήταν να είναι εδώ και να παρακολουθήσει τη συζήτηση που ακολουθεί. Και κυρίως καθώς ήταν μια πολύ σύντομη έκθεση. Ήταν εδώ πριν να φτάσετε εσείς όμως κυρία μου. Ναι, αλλά δεν ήταν εδώ για τη συζήτηση. Ναι, εδώ ήταν. Τον άκουσα που μου έκανε την εισήγησή του. Ζήτησε συγγνώμη. Ε, Συνήθω, ε, ε, ναι, ζήτησε συγγνώμη γιατί έπρεπε να φύγει. Είναι καλό άνθρωπο και το συμπαθούμε. Λοιπόν, ε, κανονισμός ε, διμερής ρήτρα διασφάλισης, εξηγητής ο κύριος Λάγκη και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Ε, αφού συζητήσαμε ήδη για το σχέδιο έκθεσής μου, υπάρχουν περαιτέρω άλλες 14 τροπολογίες που εντάσσονται στις, ε, συνάδουν με τις ιδέες μου. Πρόκειται για τέσσερα σημεία όσον αφορά το ζήτημα της ρήτρα διαφύλαξης και του μηχανισμού σταθεροποίησης. Τα εξή. Πρώτον, ε, η έκθεση της Επιτροπής και η συγκέντρωση σημαντικών δεδομένων και στοιχείων, ούτως ώστε να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιολογεί σε ποιο βαθμό ε, θα πρέπει να γίνει προσφυγή στη ρήτρα διαφύλαξης και το μηχανισμό σταθεροποίησης. Δεύτερον, ποια κριτήρια εφαρμόζονται για την αξιολόγηση και στην περίπτωση μιας ε, έρευνας προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα. Το τρίτο σημείο αφορά το πώς θα πρέπει να συμμετάσχει το Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία και το τέταρτο σημείο αφορά το μηχανισμό σταθεροποίησης της μπανάνες. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι κατατεθήσεις τροπολογίες πηγαίνουν όλες προς την ίδια κατεύθυνση όπου εγώ ίδιος ε, μπόρεσα να κάνω κάποιες προτάσεις και πολλές ε, τροπολογίες σχεδόν ταυτόσιμες. Για παράδειγμα, η 32 είναι μια συμπλήρωση, προσθήκη. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι μπορούν να ενταχθούν όλες στην έκθεση. Άρα λοιπόν τα τέσσερα αυτά σημεία έχουν επιλεγεί σωστά και τη χάνουν τη συμφωνία των ε, συναδέλφων. Ε, το μόνο το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε είναι το εξής. Υπάρχει η πρόταση να επεκταθεί η νομική βάση και το 349, όχι μόνο το 207 όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ε, δεν το έχω εντελώς ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό στο κεφάλι μου, γι' αυτό θα προσφέξω σε νομική, στη νομική υπηρεσία όσον αφορά τα δικαιώματα των παραγών μπανάνα στις εξόχως απόκεντρες ε, περιοχές. Ε, κατά πόσο λαμβάνονται αυτά τα δικαιώματα υπόψη. Ε, σχέση με την νομική βάση. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, όπως σας είπα, νομίζω ότι μπορούν να σωματωθούν όλες τις τροπολογίες και όσον αφορά την νομική βάση θα πρέπει να το δούμε εκ του σύνεγγης. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τις τροπολογίες. Η Χωσέφα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση για την, για την ίδια τροπολογία με την προηγούμενη έκθεση και αφορά το μηχανισμό σταθεροποίηση για τις μπανάνες. Ε, είπε ο κύριος Λάγκη και τον ευχαριστώ ότι οι τροπολογίες συνάδουν με την έκθεση. Περιμένουμε και την νομική έκθεση για τις άκρως μακρές περιοχές. Θέλω όμως να κάνω μια ερώτηση στην Επιτροπή που μας έδωσε κάποιες εξηγήσεις. Τι διαφορά υπάρχει μεταξύ αυτό του μηχανισμού σταθεροποίησης και της ρήτρα διασφάλισης. Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Λέτε επίσης ότι δεν μπορούν να καθοριστούν ποσοστός. Εμείς δεν μιλήσαμε για κάτι τέτοιο, αλλά για αύξηση ε, ενός συγκεκριμένου όγκου που πλήττει σοβαρά. Κάτι το οποίο θα έρετο με την ε, ρήτρα διασφάλισης. Αυτό που είπατε για το δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εσείς ε, διαφοροποιήσατε αυτό από τα εμπορικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αξιολογήσει, λέτε, γιατί δεν έχει στοιχεία για τις ποσότητες και τις ποσοστώσεις. Δεν θα πρέπει να έχει πληροφορίες κομισιών για να δει αν υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος. Αυτές οι εκθέσεις ε, αξιολόγησης είναι σημαντικές. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι μέτρο που θα οδηγεί σε αναστολή και σε διαδικασία διαβούλευσης. Ευχαριστώ η Λούση τώρα, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή κύριο Λάγκη. Θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση για την ρήτρα διασφάλιση και το μηχανισμό σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο τέφαλο της Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κολομβία και το Περού. Θέτεται, τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2020. Το Μάρτιο του 2011, ως η συγκεκριτρία του ΕΛΚΑ για τη Συμφωνία για τις Μπανάνες, στο πες του ΠΟΕ, μια έκθεση που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο, είχα τονίσει ότι ενώ προχωράμε προς μεγαλύτερη απελευθέρωση του παγκοσμίου εμπορίου στις μπανάνες. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα εξαλείψουμε ολόκληρους τομείς και βιομηχανίες που από παράδοση διδραματίζουν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο σε ευρωπαϊκές περιοχές όπως Γουαδελούπ, Μαρτινίκα, Μαδέρα, Ζόρες, ε, Κανάρια κτλ. Είναι όλες αυτές οι περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες γιατί δεν έχουν πολλές δυνατότητες διαφοροποίησης παραγωγής. Ο προτινόμενος μηχανισμός σταθεροποίησης και η ρήτρα διασφάλισης δεν νομίζω ότι είναι αρκετά αποτελεσματική και συμφωνώ με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν ότι ο μηχανισμός σταθεροποίησης δεν θα είναι αυτόματος. Η Κομισιόν θα αποφασίζει αν θα τον εφαρμόσει ή όχι. Και αυτό μπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις όπου δεν θα αρκεί η υπέρβαση του κατοφλίου για να δρομολογηθεί ο μηχανισμός διασφάλισης. Στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής Άγκρη να απευθύνουμε έκκληση στην Κομισιόν όχι μόνο να εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό μηχανισμό, αλλά να δημιουργήσει συστήματα παρακολούθησης και να παράσχει και την κατάλληλη υποστήριξη στους παραγωγούς, ώστε παράλληλα με την τάση της απελευθέρωσης του παγκοσμίου ε, εμπορίου μπανάνας, να μπορούν οι τοπικοί παραγωγοί να είναι ανταγωνιστικοί στις αγορές. Στηρίζω την θέση του εισηγητή να ενισχυθούν σημαντικά τα σχετικά μέτρα. Ευχαριστώ. Κύριος Μιούλερ από την Επιτροπή ή ο κύριος Πάρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι θα μιλήσουμε και δύο. Εγώ καταρχάς θα ήθελα να πω παράλληλα με αυτά που είπε ο κύριος Λάγκε, ότι σε σχέση με τη στρατροπολιτήση του Περού και την Κολομβία, ουσιαστικά τα σχόλιά μας είναι παρόμοια με αυτά που κάναμε πριν για την Κεντρική Αμερική. για να πετύχουμε πλήρω το στόχο που προτείνεται σε κάποιες τροπολογίε πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Τώρα υπάρχει πάλι, όπω είπα και στην προηγούμενη περίπτωση, ιδιαίτερο βάρο για τι επιχειρήσει και για την Κομισιόν με κάποιε άλλε τροπολογίε. και τώρα θα ήθελα να επεκταθώ λίγο πιο αναλυτικά. Η και η κυρία Χωσέφα Αντρέα. Αν δεν υπάρχει πληροφόρηση, πώς μπορεί η Κομισιόν να παρακολουθεί την κατάσταση και ότι υπάρχει πρόβλημα. Ε, ακούστε. Εγώ δεν μιλώ για το μηχανισμό σταθεροποίησης, αλλά για τη ρήτρα διασφάλισης. Το γενικότερο μηχανισμό διασφάλισης, όταν υπάρχει μια έρευνα, ή τέλο πάντων τα προβλέπει έρευνα κανονισμός, και αν προκύψει κάτι από την έρευνα, εφαρμόζονται κάποια μέτρα ή δεν εφαρμόζονται. Ο μηχανισμός για να συλλέξουμε πληροφορίε και να αποφασίσουμε κατά πόσον πρέπει να εγκρίνουμε αυτά τα μέτρα διασφάλισης. Προβλέπει λοιπόν ότι κάνουμε την έρευνα. Πηγαίνουμε δηλαδή στους ενδιαφορομένους και συλλέγουμε πληροφορίες. Αυτό είναι το σύστημα και αποδίδει, διότι έχει βασιστεί στο μοντέλο των υφιστάμενων εμπορικών εργαλείων. Χρησιμοποιείται μάλιστα σε καθημερινή βάση και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. για να διασκεδάσω τι ανησυχίε τη επιτροπή σα σε ό,τι αφορά την απέτηση πληροφόρηση. Ε, να σας πω ότι οι πληροφορίε πρέπει να συλλεγούν για να δούμε αν θα επιβάλλουμε μέτρα ή όχι. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου κύριο Κλάρ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι το Κοινοβούλιο θα αποφύγει να καταθέσει τροπολογίες για τον κανονισμό αυτό που θα έρχονται σε αντιπαράθεση με την ίδια την ουσία της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Γιατί αυτό μπορεί να έχει στο αποτέλεσμα την απόρριψη της Συμφωνίας από τους εταίρους μας. Όπως και για την περίπτωση του κανονισμού για την Κεντρική Αμερική. Και ο κανονισμός αυτός, κάποιες τροπολογίες που προτείνονται, είναι αντίθετες ε, με τις διατάξεις ε, της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Σε τρεις κυρίως τομείς. Πρώτον, η πρόταση ο μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες να επεκταθεί και να ισχύει και μετά το 2020 είναι κάτι που δεν προβλέπεται η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο θα συμφωνήσει ούτε το Περού, ούτε η Κολομβία. Και δεν είναι και αναγκαίο σε καμία περίπτωση, αφού ακόμη και αν εκπνεύσει το 2020 αυτός ο μηχανισμός για τις μπανάνες, έχουμε μετά τον κανονισμό, τον ευρύτερο κανονισμό διασφάλισης, στον οποίο θα εμπίπτει. Άρα οι τροπολογίες 38-39 μας δημιουργούν πρόβλημα. Δεύτερος τομέας. Αυτές οι τροπολογίες που λένε για την αυτόματη εφαρμογή του μηχανισμού σταθεροποίησης όταν φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο όγκων, 36 και 37. Όπως προείπα για την Κεντρική Αμερική και εδώ θα δημιουργηθούν με αυτές τις τροπολές σημαντικά προβλήματα. Αυτή η αυτόματη διασφάλιση είναι μια ιδέα που δεν έχουν δεχθεί οι εταίροι μας. Νομίζω πάρα πολύ δύσκολα θα το αποδεχθούν αυτό. Έχουμε διαπραγματευτεί και έχουμε συμφωνήσει έναν μηχανισμό που ναι μπορεί να επικληθεί, αλλά δεν υπάρχει αυτόματη εφαρμογή του. Τώρα, διάσταση ΠΟΕ. Έχουμε δέσμευση στο πλαίσιο του ΠΟΕ να μην επανεισαγάγουμε ποσοστώσεις για τις μπανάνες. Υπάρχει νομική υποχρέωσή μας προς αυτό. Αλλά για να γίνει αυτόματος αυτός ο μηχανισμός, όταν ε, υπάρξει ένα κατόφλι, κάποια, κάποιοι συγκεκριμένη, συγκεκριμένοι, εκεί ε, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Τρίτη, δέσμη, τρίτη τροπολογία που έρχεται σε αντιπαράθεση με τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών είναι η τροπολογία 24 που αλλάζει τους όγκους κατοφλίου με τους οποίες ενεργοποιείται ο κανονισμός. Αν δείτε την κατάσταση στο Πέρου το 2006, η διασφάλιση θα ίσχυε όταν υπήρχε εισαγωγή 82.000 τόνων μπανάνας. Ενώ η δέσμευση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Έθρας Συναλλαγών είναι 90.000 τόνοι. Άρα η τροπολογία θέλει να μειώσει ουσιαστικά τα επίπεδα, του όγκους μετά από τους οποίους αρχίζει πλέον να ενεργοποιείται η ε, μηχανισμός, αλλά αυτό δεν το έχουμε διαπραγματευτεί με τους εταίρους μας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών, γι' αυτό και θα ήθελα να σας αποθαρρύνω από το να καταθέσετε τροπολίες που με την πίσω πόρτα, από την πίσω πόρτα μάλλον, προσπαθούν να μεταβάλουν το περιεχόμενο της Συμφωνίας Ελευθερών Συναλλαγών. Καταλαβαίνουμε πόσο λεπτό και ευαίσθητο είναι το θέμα των, της μπανάνας, εμείς ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτού του θέματος, πόσο σημαντικό είναι, ιδίως για τις από απόμακρες περιφέρειες της Ένωσης, ακριβώς για αυτό το λόγο δεν απελευθερώσαμε ε, την μπανάνα. Υπάρχει δηλαδή δασμός ε, για τις μπανάνες ακόμη. Έχουμε έναν ειδικό μηχανισμό σταθεροποίησης για τις μπανάνες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα χωρίς όλες οι απαιτήσει που συνοδεύουν σε μια έρευνα για τη διασφάλιση να πρέπει να ε, τηρούνται. Έχουμε ειδικέ διατάξεις ε, για τις άκρως αποκεντρές περιφέρειες. Ε, είναι λιγότερο αυστηρή ρήτρα διασφάλιση για τις άκρως αποκεντρές περιφέρειες μεταξύ άλλων. Και όπως σας είπα, ο γενικός μηχανισμός για τη διασφάλιση μπορεί να εφαρμοστεί ανα πάσα στιγμή και πριν και μετά το 2020 και γι' αυτό να σας πω ότι όταν θα μεταρρυθμίσουμε και την... όταν μεταρρυθμίσαμε την ΚΟΑ το 2007 για τις μπανάνες, μεταξύ άλλων, η Ένωση παρέσχε πολύ σημαντική οικονομική ενίσχυση στον τομέα και συγκεκριμένα στις άκρες απόκεντρες περιφέρειες. Ε, ακριβώς επειδή ε, έπρεπε να ληφθεί υπόψη αυτή η πρόκληση για τις πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες, όπως η προκείμενη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ας ακούσουμε τον εισηγητή για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Έχετε σχόλια για το ότι κάποιες τροπολογίες, όπως λέει η Κομισιόν, δεν είναι συμβατές είτε με την ίδια την συμφωνία, είτε με τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την τροπολογία υπαριθμών 24, είναι σαφές ότι οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στους αριθμούς που αναφέρονται στη συμφωνία. Άρα θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό για τις τροπολογίες 24. Και το σκεπτικό είναι ότι η συμφωνία, έτσι όπως διαπιστώσαμε, δεν μας έχει υποβληθεί επισήμως. Και ως εκ τούτου ε, πρόκειται για μια συμφωνία που θα συμφωνήσουμε εμείς ε, το 2012 ή 2013, βάσει της οποίας ορίζεται ο όγκος. Ε, δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να έχουμε σαν βάση τον όγκο των εξαγωγών. Δεν είναι δυνατόν να ζητήσει κανείς αναδρομικά ό,τι του κατέβει. Δεν υπάρχει νομική δεσμευτικότητα στην περίπτωση αυτή. Άρα θέλουμε με τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας να οριστούν επακριβώς οι συμφωνηθήσεις ποσοστώσες. Αυτή τη στιγμή αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός. Και κάτι άλλο. Πολλές τροπολογίες που καταθέσαμε, λέει η Κομισιόν, δεν ανταποκρίνονται στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Αλλά νομίζω θα πρέπει να τις δει κανείς πιο προσεκτικά. Εάν δούμε για παράδειγμα τη Ροπολογία Παριθμών 21. Εδώ ε, δεν περιγράφεται επακριβώς ο μηχανισμός στη συμφωνία. Γι' αυτό έχουμε ένα περιθώριο ε, διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τις δεσμεύσεις μας έναντι των παραγωγών στην Ευρώπη και αντιστοίχως μπορούμε να τις προσαρμόσουμε σε μια ήπια μετάβαση προς ε, ένα ελεύθερο εμπόριο. Άρα, στην ίδια τη συμφωνία δεν ορίζει το μηχανισμός, κύριε Πρόεδρε. Άρα, έχουμε το περιθώριο να διαμορφώσουμε αυτό τον μηχανισμό και υπό την έννοια αυτή θα εξετάσουμε από νομική άποψη όλες τις τροπολογίες και θα, όπως είπα, θα αξιοποιώντας, όπως είπα, το περιθώριο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών είναι 29 Μαΐου. Περνάμε στο σημείο 10 νομοθετικό ζήτημα και αυτό, τροποποίηση του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο ειδών διπλής κρίσης με εισαγητή τον κύριο Φιέλνερ, είμαστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Να σας υπενθυμίσω εν είδης αγωγής ότι πρόσφατα επικαιροποιήθηκε αυτός ο κανονισμός σε ό,τι αφορά δηλαδή τον κατάλογο των ε, προϊόντων ε, διπλής ε, χρήσης, αλλά υπάρχουν συνέχεια αλλαγές στον κατάλογο αυτό. Γι' αυτό α, ρώτησε, ζήτησε μάλλον η Κομισιόν από τους συνομοθέτες να τη δώσουμε τη δυνατότητα μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων να μπορεί να τροποποιεί τον κατάλογο. Κύριε Φιέλνερ, έχετε το λόγο. Είστε εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα μισά που είχα να πω τα είπατε. Μου χαλάσατε την παράσταση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τεχνικά είναι τα όσα πρέπει να γίνουν και δεν νομίζω να είναι ιδιαίτερα επίμοχο. Πάντως είναι ένα σημαντικό ζήτημα παρόλα αυτά. Εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται πιο πολύ για μια προσαρμογή μας ε, στην πραγματικότητα της Λισαβόνας. Αυτό το νομοθέτημα δεν είναι κατάλληλο ή δεν ήταν κατάλληλο μέχρι να κάνει τις προτινόμενε αλλαγές η Κομισιό για την κατάσταση που έχουμε πλέον ως Κοινοβούλιο στην απόφαση. Δύο πράγματα. Πρώτον, επικαιροποίηση του καταλόγου προϊόντων που θα πρέπει να θεωρηθούν ως ήδη διπλής χρήσης. Είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο, από μια λεγόμενη πράσινη λίστα, πράσινο κατάλογο, απλουστευμένη δηλαδή διαδικασία, ε, ποιες μπορούμε να βγάλουμε από αυτόν τον κατάλογο. Είπατε λοιπόν και εσείς ότι πρέπει να γίνει αυτή η επικαιροποίηση αλλαγή. Και κάτι τέτοιο συνειδητοποίησαμε και εμείς ως κοινοβούλιο. Και το ζητήσαμε κι εμείς. Γι' αυτό και δεν, ελπίζω να δεν νομίζω να υπάρξουν ε, προβλήματα. Βέβαια, εγώ προτιμώ την επιτροπολογία από τις κατεξόδου της γιατί ε, καλό είναι να παρακολουθούμε ε, την κατάσταση και να άρουμε την εξοδότηση εάν δεν κάνει τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως εμείς επιθυμούμε. Στηρίζω την πρόταση λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι ούτε εφικτό ούτε λογικό εμεί ω νομοθέτε να είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάσουμε 200.000 σελίδε τεχνικέ προδιαγραφέ. Δεν είναι δουλειά μα αυτή. Και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Δεύτερον, όταν υπάρχει επιδείνωση σε μια χώρα, υπάρχει κάποιο ένα πρόβλημα που σημαίνει ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα πρέπει να έχει μια απλή διαδικασία για την εισαγωγή ειδών διπλής χρήσης, θα πρέπει γρήγορα να μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος αφαίρεσης απομάκρυνσης αυτής της χώρας από τον κατάλογο. Με αυτόν τον τρόπο το εγγυόμαστε και αυτό, με αυτή την πρόταση. Έχω κάποιες τροπολογίες για τη διαδικασία της επιτροπολογίας, για, τη, για το Omnibus, ε, για τα χρονοδιαγράμματα και γενικώ. Αυτές είναι οι μόνες τροπολογίες που έχω καταθέσει προς το παρόν. Καλή δουλειά από την Κομισιό κατά τα λοιπά. Thank you. Um, shadows, uh... Σας ευχαριστώ. Ισκιώδης, θέλει κανείς το λόγο. Mr. Zaradio, you are one of the shadows. So you agree entirely with... Συμφωνείτε απόλυτα με τον εισηγητή. Και εγώ το ίδιο. Μην του δίνετε θάρρο, μην του δίνετε θάρρητα. Ας, καλύτερα, καλύτερα να έχουμε λίγο ησυχία. Πλήρη συνένεση. Μπράβο. Ας ακούσουμε την Κομισιόν. Πιότρ Ριτσκόφσκι. Ο κύριος Βισκόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα θα πω, μιλήσω γιατί η εισήγηση που έκανε η ε, ήταν εξαίρετη και θα κάλυψε όλα τα στοιχεία που ήθελα και εγώ να αναφέρω. Το μόνο επιπλέον πράγμα που θέλω να πω είναι ότι είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου οι αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν ε, τη ζητά τον και τα κρατημέλη και με την έννοια ότι όλοι συνειδητοποιούν πως αυτές οι διαδικασίες ενημέρωσης των ελέγχων πρέπει να γίνουν με, με γρήγορο τρόπο ώστε οι εξαγωγείς μας να παραμείνουν ανταγωνιστικοί απέναντι στις τρίτες χώρες και έπειτα για να εξασφαλιστεί η ε, ασφάλεια μέσα στην Ένωση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και οι νομοθέτες ε, πολύ θα ανακουφιστούν να αρθεί πια αυτή η ευθύνη. Ε, ναι. Εσείς εισηγητή να κλείσετε τη συζήτηση. Μάλιστα, τέλος της συζήτησης. Ωραία, σας ευχαριστώ. Προχωράμε τώρα στην εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Της έκθεσης στις 29 Μαΐου και τότε θα εξεταστεί η έκθεση λοιπόν και στοχεύουμε να τον υιοθετήσουμε τον Ιούνιο. Ε, σημείο 11. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα και εμπορικές προοπτικές. Αυτή είναι μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ήτρε, που είναι η υπεύθυνη αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή και ο εισηγητής μας είναι ο Γιούλιου Βίνκλερ από το ΕΛΚΑ. Έχεις το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ήταν σαφές από την πρώτη αντιλαγή απόψεων ότι η Επιτροπή μας η Διεθνούς Εμπορίου καλωσορίζει αυτή την ανακοίνωση και την έμφαση που δίνεται στις εξωτερικές επιτυχίες του εμπορίου και τη διεθνοποίηση του, της διεθνοποίησης του. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, αναγνωρίζοντας τις ε, αξίες και τις θετικές πτυχές της ε, ανακοίνωσης. Καταρχήν, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης αναγνωρίζονται στην ανακοίνωση ανάλογα με το μέγεθος, τη δραστηριότητά της ή την προέλευσή της. Βέβαια, πολλές φορές έχω ήδη μιλήσει σε την Επιτροπή για το γεγονός ότι δεν είναι το ίδιο να έχουμε μια μικρομεσαία σε ένα παλιό κρατομέλο σε μια εδρεωμένη οικονομία και το ίδιο να έχουμε μικρομεσαία σε στα νέα κρατημέλη που ακόμα αγωνίζονται για να έχουν πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, για να μην πω για την εξωτερική διάσταση. Οι μικρές λοιπόν και οι μικροεπιχειρήσεις είναι πολύ διαφορετικές από τις μεσαίες και οι διεθνείς τους φιλοδοξίες φυσικά θα πρέπει να υποστηριχτούν με διαφορετικά μέσα. Το δεύτερο μου, ε, η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι έχουμε στην ανακοίνωση ε, μια επίκριση για τα τρέχοντα προγράμματα και αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η εθνικοποίηση και η πίστη στην, ε, στην επικουρικότητα είναι πολύ σημαντική. Έχουν γίνει πολλά σε κοινοτικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι συνεργασία μεταξύ υπάρχοντων μηχανισμών θα είναι πιο αποτελεσματική από το να εφεύρουμε καινούριου. Ε, Α χρησιμοποιήσουμε αυτό που έχουμε στη διάθεσή μα με πιο αποτελεσματικό τρόπο δηλαδή. Τρίτη μου παρατήρηση, συνεργασία ανάμεσα στου φορεί στι τρίτε αγορέ και στι αγορέ προτεραιότητα. Πιστεύω ότι η κατεύθυνση και τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση δεν ήταν ευπρόσδεκτα. Φυσικά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Για παράδειγμα, αν βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρή επίκριση όσον αφορά τα μοντέλα των κέντρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν, αν επιμείνουν οι επικρίσεις, φυσικά ε, θα πρέπει να τις, λάβουμε υπόψη και να ε, προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε εξωτερικές δε πολιτικές της Ένωσης κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να επεκταθούν και στις ΜΜΕ. Θα ήταν ένα ευπρόσδεκτο βήμα αυτό. Έχουμε βέβαια και κάποιες παρατηρήσεις όπου δεν έχουμε απόλυτη συμφωνία με την Κομισιόν. Να τονίσω πέντε ιδέες, πέντε σημεία που αφορούν κάποιες ε, ε, κατευθύνσεις όπου πιστεύω πως ε, το ανακοινωθέν θα πρέπει να είναι πιο άμεσο. Καταρχήν το γεγονός, και αυτό είναι επίσης μια ιδέα που αρκετές φορές έχω επαναλάβει εδώ στην Επιτροπή μας, στο παρελθόν, από τότε που το Small Business Act έχει δημοσιοποιηθεί, πρόκειται για το γεγονός ότι αν έχουμε μια χαρτογράφηση των ισιών των μηχανισμών και αν έχουμε τα αποτελέσματα αυτού, του, αυτής της χαρτογράφησης, τότε η σύνταξη νομοθετικών προτάσεων με δεσμευτικέ διατάξει για τα κράτη-μέλη θα ήταν ποτέ, πολύ αποτελεσματική, γιατί έτσι θα ανα, εναρμονίζαμε τι πολιτικέ μα προ τα προς τις ε. Βέβαια ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να εναρμονίσουμε τα συμφέροντα των κρατών μελών, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να αναλάβουμε την πολιτική δέσμευση και να πούμε ότι ναι, αυτός είναι ο τρόπος. Τώρα άμα τα κράτη-μέλη ε, δεν το δεχτούν, τουλάχιστον η δική μας Επιτροπή θα έχει πει ότι έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε, ε, να έχουμε οικονομική διακυβέρνηση, να έχουμε σχέδια για ένα σχηρό ευρώ, μελλοντική οικονομική συνοχή πολύ μεγαλύτερη και τα ε, ε, δραστήρια προγράμματα θα πρέπει να Είμαστε πολύ υποστηρικτικοί στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσει, οι οποίες ήδη είναι παρούσε ε, στις διεθνεί αγορές. Όμω ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως έχουμε χιλιάδες ακόμα ΜΜΕ που θα πρέπει να ενημερωθούν και να γνωρίσουν το γεγονός ότι μπορούν να διεθνοποιηθούν. Δηλαδή να υπάρξει μια έξυπνη ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Οι λύσεις Τη Ένωση, στον τομέα του λειτουργικού κεφαλαίου. Δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω λεπτομερώς γιατί είναι μακρά η συζήτηση. Πάντως το λειτουργικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ είναι ένα πολύ ε, σημαντικό θέμα. Μπορούμε να ακολουθήσουμε το πρότυπο της, ε, των ΙΠΑ ή άλλα, αλλά α κάνουμε κάτι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση. Τέταρτη μου παρατήρηση αφορά την ατζέντα για τις ΜΜΕ αλλά νομίζω ότι κάποια παραπάνω πράγματα θα πρέπει να κάνουμε για τις κρατικές προμήθειες. Ε, να πω τέλος ότι ο κατάλογος των αγορών προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το δούμε με πολύ πιο διεθνή τρόπο. Έχουμε χώρε στα Δυτικά Βαλκάνια, στα, ε, έχουμε τι χώρε Ανατολική Εταιρική Σχέση και δεν θα πρέπει μόνο να βλέπουμε την Κίνα ή την Ινδία καλύτερα να κοιτάμε τους πολύ κοντινούς μας γείτονες, όπου έχουμε και πολιτικά και οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα σε επίπεδο ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε επικοδομητικό διάλογο. Φυσικά και είμαι ανοιχτό για τα, τις παρατηρήσεις και ελπίζω πως τελικά θα βελτιώσουμε κάπως αυτή την ε, κοινοθέν. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας. Θα υπάρξει ένα σχόλιο στην ανακοίνωση της Επιτροπής Small Business Big World σε σχέση με την διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως μας είπε ήδη ο εισηγητής μας. Τώρα θα θέλαμε να ακούσουμε τους σκιώδεις. Ο κύριος Σούστα. Σύντομα, Πρόεδρε, να πω ότι είναι πολύ καλέ οι παρατηρήσει του εισηγητή. Όλοι γνωρίζουμε πόσο είναι σημαντικό και στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή ε, οικονομία αυτό ο τομέα είναι ένα κείμενο επί το οποίο θέλουμε να δουλέψουμε θετικά. Εκτιμώ όλου ιδιαίτερω στην παράγραφο 5 που σχετίζεται με την ανάγκη δεσμεύσεων, μάλλον δεσμεύσεων από τα κράτη-μέλη την 7 που αφορά τις μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε στρατηγικούς τομείς ιδιαίτερα για την τομέα της μεταποίησης όπου υπάρχει υψηλή προστιθέμενη αξία παράγραφος 8 για την ενιαία θηρίδα για εξαγωγών σε τοπικό επίπεδο την 10 για τις θηρίδες βοήθειας γραφή εξυπηρέτησης σε θέματα εμπορικής άμυνας και τη 14 ότι, που λέει ότι θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα οι γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητες επί τη βάση της ατζέντα των τρέχουσων διαπραγματεύσεων για εμπορικές συμφωνίες με διάφορες χώρες. Αυτό ο τομέας θα πρέπει να, να δώσουμε, μάλλον σε αυτό το τομέα, συγκεκριμένα στοιχεία. Αναθεώρηση του Small Business Act είναι βέβαια ένα δρόμο όπου θα πρέπει να το να στηρίξουμε και να στηρίξουμε τις ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές και ε, τα προβλήματα που έχουν όσον αφορά την ε, πνευματική διοκτησία, την ενεργοποίηση της ε, δικαστικής υπεράσπισης ενώπιων δικαστηρίων. Τέτοι, αυτός ο στόχος νομίζω έχει περιγραφεί ευρύτατα και θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε ίσως σε κάποιες συμπληρώσεις στην διάρκεια της εξέτασης αυτής της νομοδότησης. Ο κύριος Ντάρτμος. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα μπορούσε να είναι πολύ θετικό α, αν οι διακεκριμένοι συνάδελφοι είχαν και αυτοί λόγο για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να, κάνω, να θέσω τρία σημεία. Ο καθένας μας, λίγο πολύ ο καθένας μα είναι υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εδώ δεν υπάρχει εξαίρεση. Σχεδόν ο καθένας είναι υπέρ των χωρών μελών, εταιριών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξάγουν. Άρα λοιπόν ο καθένας είναι υπέρ του να εξάγουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, θα πρέπει να εκφράσω μια ανησυχία. Ότι, δηλαδή, ε, πίσω από όλα αυτά, όπου όλοι συμφωνούμε, αυτό το οποίο δεν θέλουμε να έχουμε είναι τη δημιουργία νέων δομών που είναι ιδιαίτερως δαπανηρές και δεν ξέρω εάν ε, έχουμε επίγνωση γεγονότος ότι τα μέλη της υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, πληρώνονται για να έχουν 7 εβδομάδες διακοπές το χρόνο. Όλοι ενδιαφερόμαστε για την αύξηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αλλά δεν είναι όμως αυτό ε, που επιθυμούν οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα εντάχει να διευκρινίσω δύο σημεία εδώ. Υπάρχει το σημείο υπαρθμών 5 που καλεί την Επιτροπή να συντάξει ένα νομοθετικό ψήφισμα με δεσμεύσεις εκ μέρους των χωρών μελών για να απλουστεύσουν όλες τις εθνικές διαδικασίες όσον αφορά την διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλα αυτά έχουν πολύ θετικά, αλλά στην πράξη αυτό που θα συμβεί είναι ότι η Επιτροπή θα παράγει 15 σελίδες νομοθετικών ε, προτάσεων που θα δημιουργήσουν περισσότερο διοικητικό άχθος στις πλάτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις χώρες μέλη και όλα αυτά ε, εξ ονόματος δίθεν της ε, απλούς, απλούστευσης. Από την άλλη, ε, καταλαβαίνω τις ανησυχίες του εισηγητού, αλλά από την άλλη η έννοια που έχετε σχετικά μιας ευρωπαϊκής οντότητας για να ξεπεράσουμε την έλλειψη προσωπικού της μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω. Ε, ξέρετε τι γίνεται. Έχετε πάει ποτέ σε καζίνο στη ζωή σας. Εάν πάτε στο καζίνο βλέπετε ότι εκεί ε, δίδονται κάποια ποσά και από την άλλη πληρώνονται κάποια ποσά, ε, τα κέρδη δηλαδή. Αλλά τελικά πληρώνουν περισσότερο οι πελάτες του καζίνο για να παίξουν από αυτό πληρώνει το καζίνο για τα κέρδη. Και αυτό συμβαίνει με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν πραγματικά είχαμε μια ευρωπαϊκή ένωση, μια ευρωπαϊκή οντότητα που να παρέχει κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήταν καλό, αλλά αυτό που, στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι οι χώρες μέλη πληρώνουν τεράστια ποσά σε μια εποχή όπου οι φορολογούμενοι στις χώρες μέλη δεν επιθυμούν διακαώς να πληρώνουν περισσότερα χρήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα υπάρξει μια τεράστια γραφοκρατία στο μέσον και μικρά πενιχρά κεφάλαια τα οποία τελικά θα διευθυνθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ ακριβώς εδράζεται η ανησυχία μου. Θα ήθελα να ακούσω την απάντηση του εισηγητού σε σχέση με αυτές τις ανησυχίες. Ευχαριστούμε. Πράγματι, το ερώτημα εδώ είναι κατά πόσο υπάρχει προσθέμενη αξία όσον αφορά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ακούσουμε τώρα τον ε, Χωσέφ Ανδρέας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η τελευταία παρένταση μας έδωσε την οπτική του γκρουπιέρι ε, σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση πραγματικά έχει μεγάλη σημασία γιατί αναφέρεται στην αύξηση ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας το 85% των θέσεων απασχόλησης προέρχονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυστυχώς δεν υποφελούνται από αυτές τις ε, δυνατότητες συντονισμού όλων αυτών των στοιχείων. Και θα πρέπει να επωφεληθούν όμως από την διεθνοποίηση των αγορών και από την αύξηση των δυνατότητων πρόσβασης στις, αγοράς, ε, στις αγορές αυτές. Ε, μέσω δημιουργίας νέων δικτύων, μέσω αύξηση της διαφάνειας της μέσω δυνατότητας πρόσβασης στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω στρατηγικής 2020. Και αυτό σημαίνει στο δυναμή με την αναζήτηση νέων τρόπων δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των ευκαιριών. Και συνεπώς η έκθεση αυτή έχει, είναι ουσιαστική όσον αφορά την αναζήτηση απασχόλησης. Και νομίζω ότι τα σχόλια μας θα πρέπει να έχουν το νόημα ενίσχυσης αυτής της έκθεσης που έχει στον πυρήνα της ακριβώς τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την πολύ ακριβή περιγραφή της κατάστασης και για τις ε, προτάσεις του. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση αυτή πηγαίνει προς την ορθή κατεύθυνση και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω όλοι μας δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να αυξήσουμε το μερίδιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ελληνικό όγκο επενδύσεων και εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες εκτός. Ιδιαίτερα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην παράγραφο 9 υπάρχει μια αναφορά για τις μικροεπιχειρήσεις που ενίοτε παραμελούνται. Και γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα στο γεγονό ότι ο κύριος συγητής κάνει αυτή τη μνήα. Επίσης πιστεύω ότι υπάρχει και μια άλλη πιο σημαντική σημείωση στην παράγραφο παριθμών 12 που έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνους από εμά που ακόμα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο κύμα διεύρυνσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσει από νέες ή μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ορισμένε φορέ βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια μνήμα που είναι σημαντική. Επίσης θα ήθελα να... Αλλά από την άλλη θα ήθελα να ομολογήσω ότι είναι ορισμένοι... υπάρχουν ορισμένοι παράγραφοι που θεωρώ ότι παρουσιάζουν κάποια προβλήματα και συμφωνώ με κάποιον από τους προλαλήσαντες ότι ιδιαίτερως η των παραγραφών 5 και 11 κατά την άποψή μου, επιδέχονται περαιτέρω διευκρινήσεων και ε, καμιά φορά οι καλές προθέσεις δεν είναι αρκετές και ορισμένες φορές ίσως οι καλές προθέσεις χρησιμοποιούνται ως ε, αυτοσκοπός για ε, επαύξηση, υπερτέρα επαύξηση του γραφειοκρατικού άχθους. Άρα λοιπόν θα πρέπει, λίγο, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην διολυσίσω το πράγμα σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά κατά βάση συμφωνώ με την έκθεση και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή και εάν υπάρχει κάτι που δημιουργεί ε, διαφωνήσεις θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Ωραία. Κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών με τον κύριο Ράμστορφ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την, πραγματικά, για την έκθεση του που πραγματικά κουρεί τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί 70% των θέσεων απασχόληση προέρχονται ακριβώς από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα έχουν ένα μερίδιο μόνο 4% όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν οι αριθμοί αυτοί περιγράφουν πολύ καλά τη δυσχερή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ιδιαιτέρως στις νέες χώρες ε, μέλη όπου δεν έχουν αρκετά κεφάλαια και όπου δεν ε, κάναμε τίποτα υπέρ αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί όταν, για παράδειγμα, πριν από μερικά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίναμε μία έκθεση για τις μικροπιστώσεις, ε, τελικά δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Και ταυτόχρονα στην Ασία και άλλες περιοχές του κόσμου έχουμε 200 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια ανθρώπους που επωφελούνται από τις μικροπιστώσεις ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκούμεθα σε μεγαλοσχήμονες εξαγγελίες ε, για το θέμα αυτό, συζητήσεις, συζητήσεις, στις επισυζητήσεων. Και θα έλεγα ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Η... Τι γίνεται με τους ανταγωνιστές, ανταγωνιστές μας. Τη είπα, ε, εγκρίνονται ε, πολλά μέτρα, για παράδειγμα το κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, για να προωθηθούν ακριβώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ενδεχομένως οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα ζητήσουν από τα μέλη της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τις υποστηρίξουν. Ναι, θα δεχθώ μια εξαίρεση και θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο των Πρασίνων, γιατί μέχρι στιγμή δεν ακούστηκαν σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία σε αυτή την γνωμοδότηση, ιδιαίτερω όσον αφορά την πτυχή τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμεί θα υποβάλουμε μια σειρά τροπολογιών σε σχέση με τον τρόπο που μπορούν να προστατευτούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον διεθνή ανταγωνισμό που, ενδεχο... που ορισμένες φορές είναι αθέμητος και τις οδηγεί σε πολλές σοβαρές δυσκολίες. Ενώ τα μέτρα αντι-dumping, το θέμα της δημόσιας αγοράς και του... της προσπάθειας ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί θεωρώ ότι η πραγματική αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τις υπερασπιστούμε από ένα θέμητο διεθνή ανταγωνισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να είμαστε πιο πειθαρχημένοι γιατί έχουμε καθυστερήσει με το χρονοδιάγραμμα. Σα ξαναλέω, 32 θέματα έχουμε στην διάταξη για τη σημερινή μας ε, συνεδρίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυριαζής, κύριος Κυριαζής. Yes, uh, thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και τους ε, βουλευτές που έκαναν πολύτιμα σχόλια. Εξετάσαμε τη γνωμοδότηση πάρα πολύ ενδελεχώς και είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος ε, για τα περισσότερα στοιχεία της ανακοίνωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της ανακοίνωσης, λαμβάνει υπόψη ε, το μέγεθος, ε, το τομέα και το, την τοποθεσία όπου είναι κατεστημένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ιδιαιτερότητες ε, που διέπουν τις πολιτικές μας ούτως ή άλλως. Ο στόχος μας, όπως προείπα στην προηγούμενη συζήτηση, δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο μηχανισμό που θα αλληλοπικαλύπτεται με ό,τι ήδη υπάρχει, αλλά ουσιαστικά ε, να έχουμε μια συγκεκριμένη προβολή για τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλες οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι ΜΜΕ, να, γνωρίσουν, να γνωρίζουν τι υπάρχει. Ναι, υπάρχουν ε, κάποιες χώρες που έχουν προγράμματα, άλλες που δεν έχουν για, την, ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να τον γνωρίζουν και για χώρες ε, που είναι γειτονικέ, αλλά και για αναπτυσσόμενες χώρες από άλλες υπήρους. Δεν ε, θα προτιμήσουμε μόνο μέτρα που ενθαρρύνουν με έψιλο να μετεγκατασταθούν σε χώρες όπως Κίνα, Ινδία ή Βραζιλία, αλλά και σε γειτονικέ χώρες, όπως είπατε, παραδείγματος χάρη χώρες της Ανατολικής γειτονίας ή χώρες των Βαλκανίων. Επίσης, σημειώσαμε ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβεί σε μια νομοθετική πρόταση για την λήψη δεσμευτικών μέτρων που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ. Εκφράσετε την άποψη ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αντιταχθούν σε κάτι τέτοιο πολλά κράτη-μέλη, θεωρώντας ότι είναι εθνικό το ζήτημα. Σημειώνουμε όμως και το πολιτικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε με την πρόταση αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα την οικονομική ενίσχυση των ΜΜΕ, θέλω να πω ότι ήδη στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα καινοτομή για το 2007-2011, 170.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποφελήθηκαν ήδη από κονδύλια του προγράμματος SIP, που γνωρίζετε ότι πλέον ε, έχει λιγότερα κονδύλια σε σχέση με άλλα ταμεία μήπω τα διαρθρωτικά. Ανάλογες πρωτοβουλίες προβλέπονται και στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 2014-2020. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για τα σχόλιά σας που είναι πολύτιμα για την υλοποίηση της ανακοίνωσης αυτής. Πρόεδρος Βίνκλερ, Βλέπετε ότι υπάρχει ευρεία στήριξη για την εκθεσή σας. Υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις. Ε, θέλετε να απαντήσετε, έχετε το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους αγαπητούς συναδέλφους για τη συζήτηση. Μια συζήτηση πολύ εστιασμένη, ακούστηκαν πολλές ε, καλές ιδέες. Να σας ευχαριστήσω για τις προτάσεις σας, για την υποστήριξη και για τις ε, επικρίσεις σας. Συμφωνώ απόλυτα, για να σας δώσω κάποια παραδείγματα, συμφωνώ απόλυτα με το ότι κανένα ευρωπαϊκό, μάλλον κανένα αμερικανικό μοντέλο δεν μπορεί ε, να αντιγραφεί όσο έχει και να ισχύσει για την Ευρώπη. Πρέπει να εξευρωπαϊστούν δηλαδή ε, τέτοια μοντέλα. Συμφωνώ επίσης ε, και με τον επικριτικό συνάδελφο αλλά και με την Επιτροπή την Ευρωπαϊκή. Φυσικά ε, και δεν εννοούσα εγώ ούτε νέους μηχανισμούς ούτε νέους θεσμούς. Έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει νέα εστίαση και νέες συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων μηχανισμών. Ε, για κάποιους δόριους ύπους ε, που μιλήσαμε. Να δώσω και εγώ ένα δεύτερο πολιτικό μήνυμα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί στο Κοινοβούλιο που ευχαρίστως θα δημιουργούσαν δούριους ύπους που τελικά θα βοηθούσαν την οικονομική διακυβέρνηση το ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι πιο συνεκτικό και ισχυρότερο. Είμαι ένας από αυτούς αγαπητοί συνάδελφοι και το παραδέχομαι. Και θα μ' άρεσε και θα ήθελα η Ευρώπη να είναι πιο συνεκτική και πιο συντονισμένη στο μέλλον. Για τα καζίνο Ο καπιταλιστικός ε, του καζίνου είναι αυτός που μας έχει φέρει σε αυτή την κρίση. Δεν μιλάω για την Ευρώπη, για την παγκόσμια οικονομία μιλάω. Αν λοιπόν μπορούμε να δώσουμε σε, αυτή, σε αυτόν τον καπιταλισμό του καζίνου μια απάντηση ευρωπαϊκή, μπορούμε να πούμε, ή τουλάχιστον εγώ μπορώ να πω, ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, έψιλον δηλαδή, που αποτελούν αντίβαρο ε, για τον αμερικανικό καπιταλισμό του καζίνου θα ήταν μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για το σχέδιο έκθεσης Βίνκλε 10 Μαΐου 6 το απόγευμα. Το ίδιο, η ίδια προθεσμία ισχύει για οποιαδήποτε τροπολογία στην, Επιτρο... στην έκθεση τη ΙΤΡΕ και για τη μηχανική πολιτική, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, έκθεση για την οποία τροπολογίες επιβάλλ... υποβάλλονται απευθείας στην ΙΤΡΕ και όχι στην ΙΝΤΑ. Παίρναμε τώρα στο σημείο 12, εμπορικές πτυχές της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Έκθεση ιδίω πρωτοβουλίας της δικής μας Επιτροπής Μίλοσλαβ Ράνσντορφ είναι ο εισηγητής. Το σχέδιο έκθεσης έχει ήδη παρουσιαστεί, είχε γίνει μια πρώτη συζήτηση και τώρα θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Πολλές τροπολογίες. ...142 τον αριθμό. Ο εισηγητής μου είπε ότι θα προτείνει αναβολή της ψηφοφορίας για την προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής μας, δηλαδή τη συνεδρίαση του Μαΐου. Και κάτι άλλο. Κοίταξα έτσι κάπως ακροθυγώς τις τροπολογίες, εκ των οποίων θεωρώ ότι αρκετές ε, δεν είναι μέσα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μας, δηλαδή εμπόριο και διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Ίσως λοιπόν αναγκαστώ να κρίνω ορισμένες από αυτές μη παραδεκτές. Και αν αυτό καταστεί αναγκαίο, θα σας ενημερώσω το συντομότερο δυνατό. Εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από τις μπανάνες ε, και άλλα κεντροαμερικανικά και λατινοαμερικανικά ζητήματα, περνάμε σε λιγότερο εύγευστα ζητήματα, βότκα, κρασιά, μπράντι κτλ. Οι εταίροι μας ε, στον τομέα αυτό της ανατολικής εταιρικής σχέσης θέλω να πω ότι είμαστε, ε, είμαι μάλλον ευγνώμων στους συναδέλφους μου οι οποίοι κατέθεσαν τις 142 τροπολογίες. Πάρα πολλέ τροπολογίες λοιπόν για αυτό το θέμα, για ε, το σχέδιο της έκθεσής μου και ελπίζω αυτό να δείχνει πόσο ζωτικό ενδιαφέρον ε, τρέφουν οι συνάδελφοι για τις εμπορικές πτυχές της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Είναι σημαντική η έκθεση γιατί καλύπτει πλήρως ε, ένα μια πολύ μεγάλη επικράτεια. Έχω μελετήσει τροπολογίες. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς και σε συνεργασία με τους αξιότιμους συναντέλφους ελπίζω να βρεθεί χώρος για συμβιβασμούς. σε αυτό το χρόνο θα προτείνω στους συναδέλφους μου να γίνει μια συνάντηση μεταξύ μας για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το ενδεχόμενο κατάθεση συμβαστικών τροπολογιών που εγώ θα υποβάλω αλλά και την όλη στρατηγική ώστε το συντομότερο δυνατόν να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ένας μεγάλος αριθμός τροπολογιών θέτει ευρύτερα ζητήματα, εργασιακά, κοινωνικά, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον κτλ. Ταυτόχρονα πρέπει να τονίσω ότι δεν μπορούν να ληφθούν όλα υπόψη. Εμείς εδώ εργαζόμαστε στο πλαίσιο της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Για παράδειγμα δηλαδή, τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να υπερβαίνουν το πεδίο αρμοθετών τη Επιτροπή μα. Αυτέ οι πτυχέ εξετάζονται σε άλλε επιτροπέ, όπω είναι η Επιτροπή ΑΦΕΤ, για παράδειγμα. Ο πρόεδρό μα, κ. Μορέιρα, σε μια συνεδρία είχε τονίσει ότι η έκθεση αυτή αφορά τι εμπορικέ πτυχέ τη ανατολική εταιρική σχέση όχι τις πτυχές που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορες χώρες της ε, ανατολικής σχέσης. Εγώ λοιπόν θα σεβαστώ την παρατήρηση αυτή του Προέδρου μας και θα συνεχίσω να επικεντρώνω τις δραστηριότητες μου και την έκθεσή μου στις εμπορικές σχέσεις με τους ανατολικούς μας εταίρους. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση των τροπολογιών, τι ζητήματα δηλαδή θέτουν και τα λοιπά Πρώτον, ένας μεγάλος αριθμός τροπολογιών αφορούν την έκθεση που το σημείο της έκθεσης αφορά την Ουκρανία που είναι ίσως το σημαντικότερο κράτος στο πλαίσιο αυτής της ανατολικής εταιρικής σχέσης με περίπου 46 εκατομμύρια κατοίκους και όπως πολύ καλά γνωρίζετε η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας ξεκίνησε να ισχύει από τις 30 Μαρτίου και αφορά μια πάρα πολύ ευρεία περιοχή. Κάποιες από τις τροπολογίες αλλά και ένα μέρος της εκθεσής μου καθίσταται ε, παροχημένο μετά από τη συμφωνία αυτή, γι' αυτό και πρέπει να γίνουν τροποποίησεις. Κάποιες τροποποίησεις επίσης αφορούν την ανατολική σκέψη Β, το recital Β, που λέει ότι θα πρέπει οι ανατολικοί εταίροι μας να έχουν την ίδια προσοχή με αυτή που δίνουμε στους εταίρους μας από τη Νότια Μεσόγειο. Και προτείνουν Διαγραφή. I not... Δεν νομίζω όμως ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ούτε θα ήταν δίκαιο προς τους ε, ανατολικούς εταίρους. Η Αραβική Άνοιξη δεν μπορεί να σημάνει αναγνώριση της ανατολικής ε, γειτονίας. Το έχουμε πει πολλές φορές και την ίδια γραμμή θα τηρήσω και στην έκθεση. Πολλές τροπολογίες έχουν κατατεθεί για το βήμα της έκθεσης που αφορεί, αφορά συγγνώμη, τη Λευκορωσία. Περισσότερες από αυτές αφορούν θέματα που δεν σχετίζονται με το εμπόριο, κυρίως ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικές υποθέσεις. Εξού και δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω. γιατί θα ακολουθήσω ε, την προσέγγιση που παρουσίασε ο πρόεδρός μας γι' αυτό το θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνω τις ε, θερμές μου ευχαριστίες προ τα σχόλια της προτάσεως, τις τροπολίε που θα καταθέσετε, που έχετε μάλλον καταθέσει και σας υπόσχομαι να σας προσκαλέσω σε το χρόνο σε μια συζήτηση για τα θέματα που ανέφερα στην ομιλία μου. Ελπίζω πολύ σύντομα να καταφέρουμε να φτάσουμε σε θετικά αποτελέσματα για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή έχουμε αργήσει ήδη 10 λεπτά για τη συνδράση των συντονιστών, πάρα πολύ σύντομα ε, να ζητήσω από όλους όσους λάβουν το λόγο να είναι πάρα πολύ σύντομοι. Δύο λεπτά ο κύριος Κιθ Τέιλορ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν σας είχα δει. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, συγγνώμη, και πρέπει να αρχίσουμε με τους ε, αντιπροέδρους, ο κύριος Ζαλεύσκη. Δεν ακούγεται ο κύριος Ζαλεύσκη. Εγώ θα μιλήσω πολωνικά. Σας ευχαριστώ. Εγώ διάβασα αυτό το κείμενο και πρέπει να σας πω ότι η εμπορική συνεργασία κυρίως ε, σε αυτές τις ε, συμφωνίες είναι, θέμα κλειδί για τις ε, χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Ε, υπάρχουν όμως κάποιες πτυχές για τις οποίες θα πρέπει να συζητήσουμε ήδη από σήμερα, διότι είναι πολύ σημαντικές και διότι όλα αυτά συνδέονται και με ορισμένα πολιτικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Γνωρίζουμε ποιε είναι οι πολιτικές, ε, τα πολιτικά κίνητρα που μας οδήγησαν ε, στην Ανατολική Συνεργασία. Υπάρχει ένα πλαίσιο, μια ιδέα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει σχέσεις ε, με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χάρη στι συμφωνίε συνεργασίας που προβλέπουν και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 ε, εμπορικές συναλλαγές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε χώρες όπως η Ουκρανία. Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε συμφωνίες σύνδεσης και άρα κατά συνέπεια και συμφωνίες ε, ελευθέρων συναλλαγών. Ε, το θέμα της σύνδεσης θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο ως εργαλείο ανταλλαγής με ε, ανταλλαγής ε, ε, εμπορικών συναλλαγών μάλλον, αλλά πρόκειται και για ένα είδος αποζημίωσης για το γεγονός ότι προσπαθούν να περάσουν σε μια μεταρρύθμιση, εκδημοκρατισμό και επικράτηση του κράτους δικαίου. Συνειδητοποιώ βέβαια ότι το διακύβημα είναι πολύ ευρύ και άρα δεν είναι μόνο η Ουκρανία που ε, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα αλλά και χώρες όπως το Αζερβαϊτζάν ή η Αρμενία δεν θα είναι σε θέση να συνάψουν ε, συμφωνίες σύνδεσης διότι η Ουκρανία σε αυτή τη φάση γνωρίζουμε ποια είναι η εξέλιξή της μέσω της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Διερωτώμε λοιπόν πως θα πρέπει να έχουμε μια στάση πιο ευέλικτη όσον αφορά το ότι συνδέουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ε, δεν λέω παρατήτω σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα πριν τα τέλη του χρόνου και στις αρχές του επόμενου, θα ήταν σκόπιμο να προβληματιστούμε για την πολιτική ανάπτυξη των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης με ε, μια πιο ευέλικτη στάση. Για υπάρχουν χώρες όπως η Γεωργία, η Μολδαβία, που είναι σε καλύτερη θέση για να συναυθεί συμφωνία ε, σύνδεσης και ίσως και συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Και έπειτα υπάρχουν και χώρες όπου έχουμε κάποια περισσότερα προβλήματα όπως ε, το Αζερβαϊτζάν, για να μην πω για την Αρμενία, την Ουκρανία για την οποία ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε πρόοδο και θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και τις άλλες χώρες με τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία ελευθερών συναλλαγών. Θα μπορούσαμε λοιπόν κατά τη γνώμη μου να είμαστε πιο ευέλικτοι και για τις εμπορικές σχέσεις με τη Λευκορωσία η οποία δυστυχώς στο εγγύς μέλλον, λόγω της κυβέρνησης που έχει, δεν θα είναι σε θέση να υπογράψει συμφωνία σύνδεσης. Κατά τη γνώμη μου, η σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας μπορεί να έχει ωφέλιμο σε επιπτώσεις για διαδικασίες που εμείς περιμένουμε από τη Λευκορωσία, όπως εξυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός. Θέλουμε να... Θα πρέπει μάλλον να ξαναδούμε λίγο τη θέση μας και τη στάση που έχουμε κρατήσει μέχρι στιγμή σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες. Και τώρα να περάσω στις τροπολογίες. Καταρχήν, Γεωργία και Μολδαβία. Ο εισηγητής λέει ότι θα πρέπει να επιτραπούν κάποιοι κάποια αγαθά από τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας. Ορισμένα από αυτά τα αγαθά θα πρέπει να ωφεληθούν από το καθεστώς ελευθέρων συναλλαγών. Μιλάει ο συγκεκριτής για αγαθά. Για μένα αυτό σημαίνει αποζημίωση ε, αυτών οι οποίοι απομόνιασαν αυτά τα εδάφη από τη Γεωργία και διαφωνώ με αυτή την ιδέα. Έπειτα, η Συμφωνία Ελευθέρων ε, Συναλλαγών δεν αφορά μόνο αγαθά, αλλά και θέματα ρυθμιστικά τα οποία μπορούν να αλλάξουν μόνο σε ε, περίπτωση που ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη επικράτεια θα είναι μέρος ε, του κράτους με το οποίο συνάπτεται η συμφωνία. Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι η Αυχαζία που κατέχεται από τη Ρωσία θα μπορούσε ποτέ να εφαρμόσει όλες αυτές τις αρχές για τις οποίες γίνεται λόγος στη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Μια άλλη πτυχή που κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο καθεστώς ελευθέρων συναλλαγών. Ένα άλλο τμήμα είναι η υπερδνηστερία. Εκείνο το κομμάτι δηλαδή της Μολδαβίας, ε, Δυστυχώ δεν μπορούμε να κάνουμε πιο εις βάθος συζήτηση, θα μπορούσαμε ακόμα πολλά να πούμε, αλλά δεδομένου ότι ο εισηγητή μα υποσχέθηκε ότι θα έχουμε μία ε, σύσκεψη, θα τα συζητήσουμε σε άλλη ευκαιρία. Τέταρτη φορά ε, που κάνουμε ανταλλαγή απόψεων έξεταση του σχεδίου έκθεσης θα πρέπει να περιοριστούμε σας παρακαλώ για τη συζήτηση των ε, τροπολογιών. Να δώσω τώρα το λόγο λοιπόν στους υπόλοιπους και οι Όδης Κούτας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ έχω υποβάλει 17 τροπολογίες σε αυτή την έκθεση. Ορισμένες είναι προτάσεις αναδιατύπωσης και δεν αφορούν την ουσία. Πάντω είναι γεγονό ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ πλήρης και καλογραμμένη. Θα ήθελα ωστόσο να επιστήσω την προσοχή στο ρόλο της ευρωπαϊκής αγοράς για τις χώρες των εταίρων μας προς Ανατολάς. Ορισμένες τροπολογίες από αυτές που έχω υποβάλει θέλουν να υπογραμμίσουν αυτή, ακριβώς, το, αυτόν ακριβώς τον ρόλο. Ήθελα μάλιστα να τονίσω και τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί βλέπω πως οι απόψεις δεν είναι και ομόφωνες για τα θέματα αυτά. Στην Επιτροπή Εμπορικών Διεθνούς Εμπορίου δεν ασχολούμαστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς όμως πολλές εκθέσεις συμπεριλαμβανομένες σε τούτες εδώ τις προηγούμενες για την Κολομβία. Ο εισηγητής μας εξέφρασε τις ανησυχίες του σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην ε, Κολομβία. Πολλέ εκθέσει όμω λαμβάνουν υπόψη και την ε, διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό ε, υποβάλλουμε τροπολογίε ή στηρίζουμε τροπολογίε που θεωρούμε χρήσιμε για τι συμφωνίε εταιρική σχέση που θέλουμε με αυτέ τι χώρε. Ε, σα ζητώ λοιπόν την υποστήριξή σα για μια τροπολογία που έχω υποβάλει, μια τροπολογία που έχω υποβάλει και για τη Συμφωνία σύνδεση που μετατράπει καθώς εγκρίθηκε σε επίσημη θέση της Κομισιόν της, ε, της Επιτροπής μας. Ε, θέλω αυτή την τροπολογία σε σχέση με τη Γεωργία, εννοώ μάλλον αυτή την τροπολογία για τη Γεωργία σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, και ελπίζω πως ε, με αυτόν τον τρόπο θα ακολουθήσουμε την ίδια λογική μέσα στις προτάσεις ε, της Επιτροπής ε, μας Διεθνούς Εμπορίου. Κάτι ακόμα που θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι στο κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη να αναφερθούν οι προτάσεις για τις πλήρεις ζώνες ελευθέρων συναλλαγών με αυτά τα κράτη των ε, ανατολικών εταίρων μας. Και για την Ουκρανία θα πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ για το ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πλειοψηφίας για τη χώρα αυτή. Δεν θα εγκρίνουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης μέχρι ότου η χώρα αυτή δεν ε, θα έχει πραγματικά μεταρρυθμίσει το... την ε, πολιτική της ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Τέιλορ. Ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν γέννη είμαστε ευτυχείς με τις πολυάριθμες ε, τροπολογίες. Ίσως να μείνει τόσο χαρούμενος ε, ο κύριος Ράνσδορφ. Αλλά νομίζω πως είναι σημαντικό να έχουμε μια στεναρή θέση και αυτές οι τροπολογίες όντως συμβάλλουν στο να έχουμε μια ε, μεγαλύτερη στεναρότητα. Τώρα, σε σχέση με την κατάσταση στη Λευκορωσία, ελπίζω πως θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε καλές συμβιβαστικές. Πιστεύω πως έχουμε, θα έχουμε, έχουμε καλή κατανόηση ε, και, και, και οπτική αυτής της πολιτικής ελευθέρων συναλλαγών Και να θυμίσω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε προσδοκίες και επιθυμίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε μόνο προς όφελος ελευθερών, του, ελευθέρου, του ελεύθερου εμπορίου. Ε, προσβλέπω λοιπόν σε διαπραγματεύσεις για επικοδομητικές ε, συμβιβαστικές τροπολογίες με τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Α ακούσουμε την πικροφτή. Να είστε σύντομος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες και δεν μας θέτουν προβλήματα. Απλώς θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό το είπε ο κ. Διαβλέσκη όσο αφορά ιδιαίτερο την ημερήσια διάταξη της βιώσιμης ανάπτυξης υποκοινωνική περιβαλλοντική έννοια, όπου οι τροπολογίες υπάρχουν τροπολογίε 60, 61 και 74. Και θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε από την πλευρά του εμπορίου. Το εμπόριο είναι δεγμένο τομέα για να προπαγανδίσει αυτές τις αξίες της χώρες αυτές. Ε, βεβαίως η συμφωνία σύνδεσης είναι ένα, μια, ένα deal, μια συμφωνία. Ε, ε και υποχρεώνουμε τις χώρες αυτές να συμμεριστούν με μας κάποιες αξίες ε, διακυβέρνησης. Και αυτό με οδηγεί στην εξή σκέψη. Υπάρχει η τροπολογία υπαρθμών 28, η οποία, την οποία θεωρώ προβληματική. Μας λέει ότι δεν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια συμφωνία σύνδεσης, θα πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη εμπορική συμφωνία. Εγώ θεωρώ ότι ε, εδώ να έχετε μία αντίφαση, γιατί μία τέτοιου είδου συμφωνία δεν ε, μπορεί να οδηγήσει στην ενσωμάτωση των δικών μας αξιών. Η τροπολογία 28 βρίσκεται σε αντίφαση με, επίσης με την τροπολογία υπαρθμών 59, η οποία αναφέρει αυτά τα οποία σας ανέπτυξα μόλις. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την τροπολογία 129 και 130, 31. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια διάμεση συμφωνία πριν από την υπογραφή του οριστικού πακέτου της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ε, και εδώ έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, γιατί ξέρετε ότι αυτό σηματοδοτεί το τέλος της ε, τεχνικής διαπραγμάτευσης. Δεν είναι δυνατόν να ισχύσει έστω και μια εμπορική συμφωνία χωρίς να προϋπάρξει μια πολιτική συμφωνία η οποία σηματοδοτείται ακριβώς με την υπογραφή της συμφωνίας. Και ο Επίτροπός μου πάντοτε υποστήριζε ότι είναι υπέρ μέτρων ενδιάμεσης συμφωνίας πριν από την ε, σύναψη της εμπορικής συμφωνίας αλλά μετά την υπογραφή και εφόσον ε, ε, έχει προηγηθεί διαβούλευση του Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να μείνουμε στην τεχνική συνθήκη και να τεθεί σε ισχύ με αυτόν τον τρόπο η εμπορική συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά τις αποσυστήσεις περιοχές, η DCFTA δεν συμπάγεται μόνο την άρση των τελωνιακών δασμών, αλλά την επέκταση των ευρωπαϊκών ε, κανόνων σε όλες τις ε, χώρες, ε, συγκεκριμένη περίπτωση τη Μολδαβία και θέλουμε να ζητήσουμε από τις χώρες αυτές να μας πούν πώς ε, προτίθενται να εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς πριν από την θέση ισχύ της DCFTA. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω αγαπητοί συνάδελφοι. Δύο από τους ε, σκιάδες συγητές συνέβαλαν καθοριστικά στις τροπολογίες αυτές και θα πρέπει να πω ότι το θέμα αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται ίσως εκ πρώτης όψης. Για παράδειγμα η Ουκρανία, η οποία είχε ε, πολλά προβλήματα ε, σε σχέση με την ε, παλαιωμένες βιομηχανίες της ε, Σοβιετικής Ένωσης και η μετάβαση προς ένα νέο τρόπο παραγωγής είναι εξαιρετικά δύσκολη αυτή τη χώρα. Πρόσφατα ακούσαμε εδώ μια παρουσίαση στην Επιτροπή Περιφερειών για μια περιοχή της Ουκρανίας και συζητήσαμε για μια εταιρεία η οποία παράγει πυράβλους ε, μεγάλου βεληνικούς. Στην επιχείρηση αυτή εργάζονται 60.000 εργαζόμενοι και τώρα ε, ε, εργάζονταν παλιά μάλλον και τώρα έχουν απομείνει μόνο 11.000 και είχαν 5 ή 6.000 μηχανικούς. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις αξίζει να διατηρηθούν, να επιβιώσουν. Και με τη μετάβαση προς νέες μορφές παραγωγής δεν είναι να επιτευχθεί χωρίς τη συνδρομή από το, απ' έξω. Χωρίς δηλαδή την ε, βοήθεια αυτών των εμπορικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ίδιο ενδεχομένω ισχύει και για τη Λευκορωσία. Με τη διαφορά ότι στη Λευκορωσία τέτοιου είδους μεγάλες επιχειρήσει σημαντικέ επιχειρήσεις δεν εγκαταλείφθηκαν και συνεχίζουν να παράγουν. Το πρόβλημα αυτό έχει ήδη τεθεί σε ένα πολιτικό πλαίσιο, αλλά γνωρίζουμε ότι η μετάβαση προς τη δημοκρατία είναι μια χρονοβόρα υπόθεση. Και καταρχήν θα έπρεπε να συμβάλλουμε στην ε, δημιουργία ενός κράτους δικαίου. Μια εύρυθμα λειτουργούσα δημοκρατία είναι μόνο το επιστέγασμα αυτών των εξελίξεων. Η βάση είναι το κράτος δικαίου. Και υπό την έννοια αυτή μπορούμε να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή ψάχνοντας ορισμένες, θα έλεγα, δυτικές ε, μορφές διοίκησης σε αυτές τις χώρες. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εισφορά σας και περιμένω με ανυπομονησία την επόμενη συνεργασία μας. Υπάρχει πρόταση κατόπιν συμφωνίας του εισηγητού και των σκιωδών να αναβληθεί η ψηφοφορία για, την, για το σχέδιο έκθεσης και των τροπολογιών και να γίνει στην προσοχή μας συνεδρίαση, δηλαδή στις 29 Μαΐου. Αυτό είναι το τέλος του δημόσιου τμήματος αυτής της συνεδρίασης και παρακαλώ όσοι δεν δικαιούνται να παραμείνουν για τη συνεδρίαση των συντονιστών, η οποία γίνεται και κλεισμένων των θερών, να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Παρακαλώ.